Να σας καλωσορίσω θερμά σε μια κοινή συνεδρίαση επιτροπών. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και η Επιτροπή Γυναικών έχουν σήμερα κοινή συνεδρίαση, τώρα το απόγευμα, και το θέμα ένα της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν έχει υποβληθεί καμία πρόταση για τροποποίηση, οπότε μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Σημείο 2 είναι έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης, της κοινή μας συνεδρίασης της 3ης Μαΐου. Τα έγγραφα υπάρχουν στους φακέλους σας. Εάν δεν καταγραφούν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Περνάμε κατευθείαν στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης. Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Προστασία θυμάτων της βίας. Και το θέμα ε, ε, συμπεριλαμβάνει και την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών Γι' αυτό το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα και των δύο επιτροπών μας, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και της Επιτροπής ΦΕΜ, της Επιτροπής Γυναικών. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε στενά. με βάση τον κανόνα υπαριθμών 51. 51. Γι' αυτό έχουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Λίμπε, που θα είναι και συμπρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής μας. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι οι δύο επιτροπές μας μαζί έχουν ζητήσει γνωμοδότηση από τη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης. Να σας θυμίσω επίσης ότι είχαμε δύο κοινέ συνεδριάσεις στις 3 Μαΐου και την 1η Ιουνίου. Δώσαμε στους δύο εισηγητές τότε τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη γνωμοδότηση και δώσαμε και τη δυνατότητα στους βουλευτές να ακούσουν τις θέσεις της Ισπανικής Προεδρίας και της Κομισιόν. έγινε επίσης παρουσίαση από τη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου σχετικά με τη θέση τους για τα θέματα που τους ρωτήσαμε. Θα ήθελα επίσης να σας θυμίσω ότι υπάρχει γραπτή γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Υπάρχει στους φακέλους σας. Το Υπουργικό Συμβούλιο συζήτησε την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασία στη συνεδρίαση του την 3η Ιουνίου. Έχουμε θέσει προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών 10 Ιουνίου, αλλά κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των εισηγητών αποφασίσαμε να ε, αναβάλουμε την ημερομηνία αυτή, να παραδίνουμε την προθεσμία. Σήμερα στόχος λοιπόν είναι να, γίνουν, να γίνει περαιτέρω συζήτηση της έκθεσης, ιδιαίτερα υπό το των απόψεων που έχουμε λάβει από την νομική υπηρεσία και μετά και υπό το φως της συζήτησης που έχει γίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Υπουργών. Εάν δεν έχει να προσθέσει κάτι ο πρόεδρος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους δύο εισηγητές μας, στις δύο εισηγητρίες μας, να δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Χιμένες από την ε, Επιτροπή Γυναικών. Παρακαλώ. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημερίζω τις κυρίες και τους κυρίους. Όπως είπε η πρόεδρος Βένσον λοιπόν, θα συνεχίσουμε σήμερα τη συζήτηση της απόφασης αυτής της Ένωσης για την προστασία των θυμάτων. Ξέρετε ότι ο δρόμος υπήρξε δύσκολος. Πολλαπλή φραγμή και εμπόδια. Ξέρουμε ότι το, ένα τέτοιο σύστημα προστασίας προϋπήρχε και έχουμε εδώ εκπροσώπους της Κομισιόν και του Συμβουλίου και μπορούμε αν χρειαστεί να τους ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε. Γνωρίζουμε πάντως όλοι και όλες ότι αυτό που ζητούν τα θύματα κυρίως είναι συνεργασία. Διότι κυρίες και κύριοι μου τα θύματα δεν καταλαβαίνουν τις μικροαντιζηλίες των θεσμικών οργάνων και τα προβλήματα των δικαιοδοσιών τα θύματα θέλουν ένα χώρο ασφάλειας και ελευθερίας. Όπως εξάλλου αναφέρεται και στο πρόγραμμα της Στοχόλμης. Ο στόχος λοιπόν είναι καλύτερη προστασία των θυμάτων και αυτό μας ενώνει Επιτροπή Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε να εγκρίνουμε τη δημιουργία ενός τέτοιου ευρωπαϊκού συστήματος και αύριο που λέει ο λόγος θα συνεχίσουμε με οτιδήποτε άλλες πρωτοβουλίες υποβάλλει η Κομισιόν η οποία υποσχέθηκε τέτοιες πρωτοβουλίες το 2011. Σήμερα λοιπόν, σήμερα τώρα θα ήθελα να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό το θέμα των θυμάτων στην Ένωση γιατί έχω, με αυτούς έχω αναλάβει δεσμεύσεις. Ξέρω ότι υπάρχουν όρια στις δικαιοδοσίες και των χωρών και της Κομισιόν αλλά εδώ τα θύματα δεν έχουν καμιά αμφιβολία, χρειάζεται συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων. Θα ήθελα και το επαναλαμβάνω να χορηγήσουμε στα θύματα ένα πραγματικό χώρο ασφάλειας και ελευθερίας στην Ένωση. Γιατί πρόκειται για θεμελιώδες δικαίωμα. Οποιοδήποτε πολίτης και κάτοικος της Ένωσης πρέπει να το έχει. Χρειάζεται λοιπόν ένας καλύτερος καθορισμός του περιεχομένου της ενίας αυτής του χώρου ελευθερίας και ασφαλείας. Γιατί νομίζω ότι δεν επιδείξαμε αρκετή φιλοδοξία κατά τη συγγραφή του προγράμματος της Στοκχόλμης. Μιλήσαμε για θύματα αλλά όχι για όλα, για όλες τις περιπτώσεις. Και ίσως τώρα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε, να συμπληρώσουμε, γιατί πολλά θύματα στην Ευρώπη χρήζουν προστασίας. Και θέλω εδώ να επιδείξουμε την φιλοδοξία που μας έλειψε μέχρι τώρα. Ελπίζω να δεχτείτε αυτά που προτείνω ώστε να χορηγηθεί βοήθεια σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Απευθύνομαι ιδιαίτερα στις γυναίκες που υπομένουν συζυγική και άλλη βία σε όλες τις χώρες και στην Ισπανία, ιδιαίτερα στην περιοχή μου την Ανταλουσία. Πολλές γυναίκες, όχι μόνο γυναίκες αλλά και πολλές γυναίκες ε, ε, απειλούνται ως προς την ασφάλεια και την ελευθερία τους. Υπάρχει οργανωμένο έγκλημα, μαφία, δουλεμπόριο κτλ. Υπάρχουν βέβαια οδηγίες σχετικές, υπάρχουν, το ξέρω. Ίσως χρειαστεί να συγγράψουμε και άλλες στο μέλλον, αλλά αυτό δεν εμποδίζει να αποφασίσουμε ήδη από σήμερα με τις υπάρχουσες το σύστημα προστασίας των θυμάτων που μας χρειάζονται. Δεν θέλω να έχω παροπίδες και μονολυθικές απόψεις, αλλά επαναλαμβάνω ότι θέλω να χορηγηθεί βοήθεια σε, όλα, σε όλες τις κατηγορίες θυμάτων για να γνωρίζουμε και εμείς πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Θα ακούσουμε τι έχει να μας πει το Συμβούλιο και η Επιτροπή, καθώς και όλους τους συναδέλφους που θα θελήσουν να μιλήσουν. Στην έκθεση αυτή, στη δική μου δηλαδή, για να τη συγγράψω προσπάθησα να έρθω σε επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους όσο το δυνατόν περισσότερους γιατί πιστεύω ότι όσο περισσότερους ακούσουμε τόσο μεγαλύτερο όφελος θα έχουμε στα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε. Το πρόβλημα δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην άκρη για να περιμένουμε. Χρειάζεται κάτι αμέσως, άμεσα για να μπορέσουν τα θύματα να υποφεληθούν. και όχι να έχουμε εδώ ένα εμπορικό επιχείρημα για τους εκλογείς μας. Ευχαριστώ κυρία Χιμένες. Δίνω το λόγο στην κυρία Ρομέρο για να ακούσουμε τις απόψεις της. Παρακαλώ κυρία Ρομέρο. Gracias, Presidenta. Ευχαριστώ. Το Συμβούλιο επρόκειτο να συναντηθεί στις 4 Ιουνίου για να συζητήσει για την κατάσταση των θυμάτων. Ένας βούλγαρος δημοσιογράφος, μία βούλγαρη, βουλγάρα δημοσιογράφος ε, δολοφονήθηκε. και κάποιος εμφανίστηκε στην αστυνομία του Λουξεμβούργου για να καταγγείλει ότι είχε δολοφονηθεί η γυναίκα του. Αυτή η μήνυση πέρασε απαρατήρητη. Κανείς δεν την είδε, ούτε και εμείς την είδαμε. Αλλά τα άτομα που έχουν, μόνο τα άτομα που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση ενημερώθηκαν. Και καθώς η αστυνομία του Λουξεμβούργου συνεργάστηκε με την αστυνομία των ε, Βρύξελων ε, για να τιμωρηθεί ο ένοχος του εγκλήματος αυτού, δεν υπήρξε καμία συνεργασία και δεν υπάρχει γενικά συνεργασία μεταξύ τέτοιων αστυνομικών δυνάμεων για την πρόληψη αυτών των ε, εγκλημάτων. Ε, τα άτομα αυτού του επαγγέλματος στην Βουλγαρία προστατεύονται. Η κυρία αυτή, η δημοσιογράφος αυτή, είχε καταγγείλει την συμπεριφορά αυτή που στρεφόταν εναντίον της και είχε προσπαθήσει να ζητήσει βοήθεια και στις Βρυξέλλες αλλά δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι συνέβη. Δεν έχουμε, όπως δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για ένα μεγάλο αριθμό τέτοιων εγκλημάτων, γιατί ο αριθμός των εγκλημάτων αυτών είναι στην ουσία άγνωστος. Στη χώρα μου ο κόσμος έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί τα πράγματα αυτά. Κάθε φορά που υπάρχει ένα περιστατικό βίας, κάθε φορά που υπάρχει ένα περιστατικό ε, δολοφονίας οι αρχές ε, επιδεικνύουν όλο και μεγαλύτερη προσοχή. Οι γείτονες δείχνουν όλο και μεγαλύτερη προσοχή και υπάρχει και ένα σύστημα καταγγελίας. Δυστυχώς στη Βρυξέλλες δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και η δολοφονία αυτή πέρασε απαρατήρητη. Ειλικρινά πιστεύω ότι αυτού του τύπου οι βιοπραγίες είναι πολύ τραγικές και δεν έχουμε στοιχεία στην Ευρώπη. Όποιος λέει ότι δεν είναι απαραίτητη η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας ε, θα πρέπει να δει αυτή την κατάσταση. Είναι απαραίτητη. Ακριβώς ε, θα δούμε ότι θα είναι απαραίτητη όταν δούμε τους αριθμούς και τα στοιχεία. Αυτό το έγκλημα συνήθως διαπράτεται στο σκοτάδι κυριολεκτικά και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μπορέσουν οι αρχές να το προλάβουν σε γενικές γραμμές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια από την Επιτροπή Γυναικών, γιατί εδώ καταλήγουμε σε κοινέ θέσεις και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συντάκτες των τροπολογιών. Είναι πολύ περίπλοκο το όλο ζήτημα. Ε, και ήταν δύσκολη και η τήρηση των προθεσμιών για την υποβολή των τροπολογιών. Ο εισηγητής από το ΕΛΚ θα ήθελε να αναβάλει, να παρατείνει την ε, προθεσμία υποβολής των τροπολογιών. Εγώ νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτή την, την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας, αλλά χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση να επιτευχθεί. Ε, συχνά τα επιχειρήματα που προβάλλονται είναι έολα, ε, έολα γιατί υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη για μια ευρωπαϊκή εντολή προστασίας. Μα ακριβώς δεν μπορείς να ξέρεις τι ανάγκες υπάρχουν όταν δεν ξέρεις τα στοιχεία και τους αριθμούς, όταν όλες οι σχετικές πληροφορίες ε, είναι στο σκοτάδι, όταν έχουμε τόσες ε, αλληλοεπικαλύψεις, ε, έχουμε τόσες αντιμαχόμενες απόψεις για την νομική βάση. Ε, και υπάρχει και το επιχείρημα ότι μέσα σε όλο αυτό τον κυκαιώνα τίποτα δεν θα είναι αποτελεσματικό. Ε, ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε σε πέρα αυτό όσο το δυνατόν πιο σύντομα και πιστεύω πως υπάρχει πολιτική βούληση για την υλοποίησή του. Επίσης, όταν μιλούμε για αυτήν την ε, δευτερεύουσα θυματοποίηση, η δευτερεύουσα θυματοποίηση λέγεται ότι υπάρχει όταν μετακινείται το θύμα. Εγώ πιστεύω ότι η προστασία πρέπει να είναι κάτι που ακολουθεί το θύμα και να μετακινείται μαζί με το θύμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος καλύτερος τρόπος. Όταν ενεργοποιείται ένας τέτοιος μηχανισμός, όταν δημιουργείται ένας τέτοιος μηχανισμός, θέλουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση και πρέπει να υπάρχει μία αρχή σε κάθε κράτος μέλος που να είναι η δουλειά του αυτό. Δεν είναι ανάγκη να είναι ακριβώς το ίδιο ή να είναι εντελώς ομογενοποιημένη η κατάσταση, αλλά κάθε κράτος πρέπει να έχει ένα αντίστοιχο νομικό σύστημα. Και δεν μιλούμε για νομική εναρμόνιση, εδώ μιλούμε για την εναρμόνιση ενός μηχανισμού, ο οποίος θα μπορεί να πυροδοτείται με τον ίδιο τρόπο και στον οποίο θα μπορεί να προσφεύγει ένα θύμα, το θύμα, σε οποιοδήποτε κράτο μέλος και αν βρεθεί. Είναι ένα, μέτρο προφυλακτικό, δεν είναι ένα μέτρο το οποίο έχει να κάνει με την ποινική δίωξη ή με την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων. Πρέπει να είναι ένας ταχύστατα κινούμενος μηχανισμός. Ακόμη δεν έχουμε έναν ορισμό ε, στην Ευρώπη ε, για την περιγραφή των αδικημάτων. Μιλούμε για την διακίνηση των ανθρώπινων όντων στην Ευρώπη, αλλά δεν έχουμε ενσκύψει στη βία. Μερικά κράτη-μέλη έχουν σχετικές διατάξεις, ας πούμε η Αυστρία έχει. Ε, συνεχιζόμενη βία, απειλές, σοβαρή βλάβη, ε, σεξουαλική βία, βιασμός, υπάρχουν όλοι αυτοί οι νομικοί ορισμοί, όλα αυτά τα αδικήματα. Πιστεύω ότι κάθε κράτος μέλος ανταποκρίνεται στα πράγματα αυτά. Σίγουρα κάτι υπάρχει σε κάθε κράτος μέλος για την αντιμετώπιση, για την ε, υλοποίηση ενός τέτοιου ευρωπαϊκού εντάλματος προστασίας, ενός ευρωπαϊκού, μιας ευρωπαϊκής εντολής προστασίας. Όποιος υφίσταται βιοπραγίες τέτοιου είδους θα πρέπει να μπορεί να απευθυνθεί στο σύστημα. Θα ήθελα να ξέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς το βλέπει αυτό. Έχει κάνει κάποια μελέτη επιπτώσεων. Τι έχει μελετήσει αυτή η μελέτη, το, την οικονομική επίπτωση, τι είδους επιπτώσεις θα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν αυτές οι μελέτες επιπτώσεων, οι οποίες θα πρέπει να προηγούνται των οδηγιών, έτσι δεν είναι. Υπάρχει κάτι που εξελίσσεται παράλληλα με τη δική μας δουλειά για την οδηγία εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω, θα πρέπει ίσως να βελτιωθεί όλη η διαδικασία. Να βελτιωθεί και η οδηγία μας. Η γενική σκέψη που υπάρχει πίσω από αυτήν. Ε, όταν θα παρουσιάσετε το σχέδιο οδηγίας ε, για την ε, βία, θα πρέπει να μπορείτε κάπως να τη στηρίξετε. Όσο δεν υπάρχει ένας ορισμός του αδικήματος, θα συνεχίζονται οι επιθέσεις, οι γυναίκες θα πεθαίνουν και πραγματικά έχουμε καθήκον να κάνουμε κάτι, να κάνουμε κάτι πραγματικό. Δεν μπορούμε να νύπτουμε τα σχήρας μας αφού έχουν τελεστεί τα εγκλήματα. Διαφορετικά θα δούμε και άλλες δολοφονίες σαν αυτές της Διάννα Παρακαδόβα, της Βουλγάρας δημοσιογράφου. Και ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε είναι να εγκαθιδρύσουμε μια διαδικασία σαν αυτή για την οποία μιλούμε τώρα και νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το σκεφτεί, να το εξετάσει εμείς είμαστε διατεθειμένοι και ανοιχτοί να ακούσουμε οποιαδήποτε νομική γνωμοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας έχει παρουσιάσει κάποια νομική ε, γνωμοδότηση. Ε, ίσως μπορείτε να έρθετε και να κάνετε αυτό που δεν έκανε το Συμβούλιο ή αυτό που δεν έχει κάνει το Κοινοβούλιο. Να συμβάλλετε, να προσθέσετε κάτι marcha un mecanismo que se nos está revelando como urgente. Gracias. Πρέπει λοιπόν να στηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός και με μεγάλη επιτακτικότητα. Κυρία Ρομέρο, σας ευχαριστώ θερμά. Ακούσαμε ένα παράδειγμα βίας, η οποία δυστυχώς όμως είναι ε, πολύ συνήθις και στόχος της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προλάβουμε αυτά τα απέσια εγκλήματα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέρφους για να ακούσουμε τις απόψεις τους. Το λόγο έχουν οι βουλευτές. Ε, ε, να δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Μορέν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι το κείμενο αλλά και το ίδιο το θέμα μας αναγκάζει όλους να θυμηθούμε τις δεσμεύσεις μας και τις ευθύνες μας. Πρέπει όλοι να ενδιαφερθούμε για αυτό το θέμα που είναι τεράστια σημασίας για την κοινωνία μας και παρόλα αυτά πολύ δύσκολο να το χειριστούμε. Το μεγαλύτερο όφελος που θα μπορούσαμε να έχουμε από αυτή την δουλειά, από την έκθεση δηλαδή, θα ήταν να δημιουργήσουμε μια συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι υπάρχει αυτή η βία γιατί συχνά είναι κάτι που κρύβεται ή που είναι άγνωστο. Πρέπει δηλαδή να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι πρόκειται για πρόβλημα που βρίσκεται σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Δεν υπάρχει κοινωνική ομάδα που να είναι ελεύθερη αυτού του προβλήματος της βίας. Και δεν πρόκειται μόνο για τους ασθενέστερους οικονομικά, για τους λιγότερο προνομιούχους, ούτε για τους πιο ηλικιωμένους, ούτε για τους πιο νέους, ούτε για τους πιο απομακρυσμένους από το κέντρο των πόλεων. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία και μπροστά σε αυτό το πρόβλημα λοιπόν έχουμε την ευθύνη και την υποχρέωση να έχουμε κάποια ανταπόκριση, να δώσουμε κάποια γρήγορη απάντηση. Θα ήθελα λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι να στηρίξουν τη δουλειά της κυρίας Χιμένες και της κυρίας Ρομέρο γιατί είναι, επαναλαμβάνω, υποχρέωσή μας να καταλήξουμε κάπου για να βοηθήσουμε τα θύματα. Δεύτερον, μερικά από αυτά τα θύματα είναι ιδιαίτερα νεαρά άτομα. Σωστό είναι ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα και δολοφονίες προσωπικότητων αλλά πρέπει επίσης να μην ξεχνάμε, δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι στη ζωή μας όλες μας και όλοι μας έχουμε συναντήσει και νεαρά άτομα ως θύματα, νεωρότερα των 10 ετών μάλιστα. Και αυτό μας υποχρεώνει να είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί και δραστήριοι. Τρίτον, η δυσκολία της αντιμετώπισης του προβλήματος δεν έγκυται μόνο στο να καταλήξουμε σε συμφωνία μεταξύ 27 χωρών που να αναλάβουν το πρόβλημα αυτό, αλλά έγκυται και στο ότι πρέπει το πρόβλημα αυτό να το αποκαλύψουμε κανονικά, γιατί πολλές φορές τα θύματα είναι μόνα τους και κρύβουν τι τους συνέβη. Ξέρουμε καλά γενικότερα ότι υπάρχει το πρόβλημα, αλλά πρέπει να δοθεί ο λόγος στα θύματα τα ίδια για να μπορέσουμε να τα προωθήσουμε και να τα προασπίσουμε καλύτερα. Τέλος, πρέπει να είμαστε πολύ αποτελεσματικότεροι. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει συντονισμός μιας ευνοσιακής δράσης μεταξύ και των 27 χωρών αν δεν καταφέρουμε κάτι τέτοιο σύντομα, ένα συντονισμό τέτοιου επίπεδου δηλαδή ώστε να ώστε ο ίδιος ο πόνος του θύματος που χρειάζεται για να αποκαλυφθεί κάτι σε κάποια χώρα να μην πρέπει να διπλασιαστεί και σε άλλη χώρα. Αλλιώς θα ήταν δικό μας το φταίξιμο. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα βασικό πρόβλημα ισότητας και προστασίας των πολιτών. Στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση λοιπόν πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί σε όλες τις πτυχές και ηλικίες της κοινωνίας και για τις γυναίκες αλλά και για το σύνολο των πολιτών. Αν η Επιτροπή Γυναικών μπορέσει να τύχει της υποστήριξης και της Επιτροπής ΕΛΕΦ τότε θα ήταν κάτι πολύ θετικό αυτό. Ευχαριστώ κυρία Μωρίν. Η κυρία Πιλπάου είναι η επόμενη ομιλήτρια. Sí, muchas gracias, Presidenta. Y muchas gracias a las ponentes por el esfuerzo que están realizando. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους, τις συζητήσεις για τις προσπάθειές τους να προωθήσουν το θέμα αυτό. Νομίζω ότι όλοι στην αίθουσα και ότι όλοι όσοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά σε θεσμικό επίπεδο θέλουν να προστατεύσουν τα θύματα της φυλετικής βίας ε, πολύ συχνά εντός της οικογένειας. Ε, συχνά ξεχνάμε τα πολύ νέα κορίτσια που πέφτουν θύματα βίας. Τα τελευταία γεγονότα που σημείωσα εγώ, είδαμε μία υπόθεση όπου μία γυναίκα αλλά και τα παιδιά της ταυτόχρονα ήταν θύματα βίας. Στον 21ο αιώνα λοιπόν δεν έχουμε την ίδια κοινωνική δομή ζευγαριών που είχαμε στο παρελθόν. Προτιμώ λοιπόν να ε, μιλώ για τα πρόσωπα που ήταν ε, θύματα ε, βίας. 18 τροπολογίες θα υποβάλω για να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την διπλή θυματοποίηση γυναικών στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τις διαδικασίες συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών. Δεν θα πρέπει δηλαδή να αναγκάζουμε τις γυναίκες να έχουν κάποιο επιπλέον κόστος για, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας για να, ε, θα πρέπει να προωθήσουμε την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών, θα πρέπει να κατακτήσουμε νέες διαδικασίες ε, για να βελτιώσουμε την προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά είναι τα κίνητρα για τις 18 τροπολογίες μου. Η ερώτησή μου είναι πότε έχει μεταφερθεί η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Στις συνεδριάσεις που είχαμε, είπα ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για να υπάρξει ανάλυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να εξεταστούν τα συστήματα που έχουμε στα 27 κράτη-μέλη. Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να γίνει ε, αν θέλουμε να εγκρίνουμε μια, ένα σύστημα με τα χαρακτηριστικά αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια διαδικασία δικαστικής αναγνώρισης. Πώς μπορεί να γίνει αυτό σε χώρες που δεν έχουν κάτι τέτοιο. Μπορεί ε, οι διαδικασίες μας ε, να είναι σύμβατες με κάποια νομικά συστήματα. Θα ήθελα πολύ να γνωρίζω ποια είναι τα αποτελέσματα. Έχουμε κάποια σχετική έκθεση και, και μία σκέψη. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία μας κατά της βίας ε, δεν βοηθάει το γόητρό μας ως θεσμικό όργανο, διότι Προσπαθούμε να προστατεύσουμε κάποιους ανθρώπους, αλλά ε, έχει γίνει αντικείμενο διαμάχης μεταξύ των θεσμικών οργάνων και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν σε αυτό και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δίνουμε αυτή την εντύπωση. Αυτή είναι η σκέψη που θα ήθελα να εξετάσουμε και θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν σε τι βαθμό θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ό,τι υιοθετήσουμε στα πλαίσια του Κοινοβουλίου. Τι είναι εφικτό μέχρι το 2011. Είναι δυνατόν ή όχι να μοιραστείτε μαζί μας σε κάποιες από τις πληροφορίες που αναλύετε και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ή όχι. Ποια είναι τα αποτελέσματα της μελέτης σας. Μιλήσατε για νομικά προβλήματα. Εγώ δεν το έχω δει το πρόβλημα αυτό. Εμείς οι νομοθέτες είμαστε οι άνθρωποι που τροποποιούμε συνεχώς τους νόμους ε, για να ευθυγραμμίζονται με την πραγματικότητα. Νομικό, το νομικό πρόβλημα λοιπόν δεν είναι δικό μας πρόβλημα, διότι μπορούμε όπως και για τόσα άλλα θέματα να κάνουμε τις νομικές προσαρμογές που είναι απαραίτητες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό είτε στη σημερινή μας συνεδρίαση είτε στην επόμενη. Ρεαλιστικά, πού θα μπορέσουμε να φτάσουμε, μέχρι πού. Σημασία δεν έχει το πώς. Πολλή δουλειά γίνεται ταυτόχρονα και αλλιώς κινδυνεύουμε να φτάσουμε το 2011 με νέα πρόταση με αποτέλεσμα ό,τι κάνουμε φέτος να είναι σπατάλη χρόνου. Μπορεί να μας εκπλήξετε, να μας υποβάλλετε κάτι νέο, αλλά ρεαλιστικά, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, μέχρι πού μπορούμε να προχωρήσουμε αυτή τη στιγμή η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα πρέπει να αναλύσουν ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει κάτι που να μπορούμε να κάνουμε, κάποια βιώσιμη λύση. Ε, αν όχι, πείτε μας όχι, να μην σπαταλάμε το χρόνο μας. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να συνεργαστούμε, να εγκρίνουμε με τη μεγαλύτερη βάση ε, συνένεσης ε, να υιοθετήσουμε κάτι που να μπορεί να βοηθήσει του ανθρώπου αυτού. Δώστε μα λοιπόν μια σαφή διαδικασία, σαφείς προθεσμίε ε, και να δώσουμε μια πιο σοβαρή εντύπωση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Να δείξουμε ότι δεν σπαταλάμε χρόνο σε μια σοβαρή υπόθεση. Ευχαριστώ η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ. άργησα λίγο. Μπορεί ήδη να έχει απαντηθεί η ερώτησή μου. Αυτό που θα ήθελα όμως ε, θα ήταν να έχω κάποιο είδους επιβεβαίωση ή διευκρίνηση σχετικά με την κατάσταση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου. Θα ήμουν πολύ περίεργη να μάθω ποια είναι η απόφαση της εισηγήτριας να εγκρίνουμε την έκθεση αυτή και να θεωρήσουμε νομική μας βάση το 82.1 ή το 81α. Ποια θα πρέπει να είναι η νομική μας βάση. Θα ήθελα επίσης να ξέρω αν εκλάβουμε ως νομική βάση το 82.1, μιλάμε για το ποινικό δίκαιο, το οποίο θα εφαρμόζεται για την ε, έκδοση Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας. Τι θα ισχύει ε, τότε για το άρθρο 81α, ότι οι σχετικές προτάσεις έχουν γίνει θα πρέπει να ανακληθούν. Και τι θα γίνει εάν υιοθετήσουμε ένα νομοθέτημα το οποίο να περιέχει αντιφάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η θέση της Κομισιόν για το θέμα αυτό, προτού να προχωρήσουμε τη συζήτηση, διότι νομίζω ότι έχουν, έχει τεθεί μια σειρά ερωτημάτων για τα οποία είναι σημαντικό να ακούσουμε τη θέση της Κομισιόν προτού να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ. Δίνω το λόγο στην κυρία Κώστα. Παρακαλώ. Ehm, Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και τις δύο εισηγήτριες. Και θα ήθελα να πω στην κυρία Χιμένες ότι όλοι έχουμε την πρόθεση να είμαστε πολύ φιλόδοξοι με το κείμενο αυτό και να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία στα θύματα αυτών των ε, διώξεων που μπορούν να φτάσουν μέχρι και στην ανθρωποκτονία και το θάνατο. Ε, πρέπει όμως να κατανοήσουμε υπό ποια έννοια είμαστε φιλόδοξοι. Εγώ νομίζω ότι ευκταίο είναι φυσικά να υπάρξει μια προοπτική και ίσως και μια ευρύτερη οδηγία για όλα τα θύματα της βίας. Σας υπενθυμίζω ότι εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή πάνω σε πολλά κείμενα. Για παράδειγμα έχουμε ένα σημαντικό κείμενο για τη διακίνηση των ανθρώπινων όντων που είναι ένα ειδικότερο ζήτημα. Ε, εδώ έχουμε μια πρωτοβουλία 12 κρατών μελών. Σίγουρα λοιπόν υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που νιώθουν επίγον να παρέμβουν στον τομέα, στο ζήτημα αυτό. Και αυτό δείχνει ότι το, το Κοινοβούλιο συμμετέχει. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όμως ποιους τύπους θυμάτων, ποιες κατηγορίες θυμάτων θέλουμε να προφυλάξουμε. Ε, είναι μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Είναι άτομα τα οποία έχουν ήδη πετύχει την έκδοση κάποιας εντολής προστασίας στη δική τους χώρα. Και ανεξάρτητα από την νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους, θα πρέπει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων στο έδαφος της. Άρα έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων μπροστά μας που θέλουμε να προστατεύσουμε. Εντάξει, θα ήταν πολύ ευκταίο να έχουμε να στοχεύσουμε σε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Πάντοτε υπάρχουν περισσότερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί η φιλοδοξία πρέπει να βρίσκεται στην, ε, να εκφράζεται στην νομική βάση που θα επιλέξουμε ως βάση αυτού του νομοθετήματος. Ε, εδώ επιδεικνύεται μια πολύ μεγάλη καινοτομία, μια πολύ μεγάλη ε, πρωτοπόρα έτσι προσέγγιση. Και συγχαίρω τη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου που επέλεξε τη συγκεκριμένη νομική βάση στη νομική της γνωμοδότηση, το 82.1 συγκεκριμένα. Αλλά υπάρχει και μια πιο φιλόδοξη νομική βάση και συγκεκριμένα το άρθρο 3 το οποίο δεν επιτρέπει αλλά υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια άτομα τα οποία χρήζουν και αξίζουν μια συγκεκριμένη προστασία. Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλη διασαφήνιση και όχι, δεν μου φαίνεται ότι προκαλεί σύγχυση. Το άρθρο 3, όπως λέει η γνωμοδότηση της, Επιτροπής, της Νομικής Επιτροπής, ε, προσδίδει μια διαφορετική φύση στην προσπάθειά μας. Ε, εκφράζει ένα άλμα, γιατί είναι αδιάφορο ποια αρχή, αν ήταν αστική, διοικητική ή ποινική, που εξέδωσε αυτή την εντολή προστασίας. Η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας θα προστατεύει όλα τα άτομα που έχουν επιτύχει την έκδοση μιας τέτοιας απόφασης στη χώρα τους. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να καλύψουμε ένα ευρύτερο φάσμα αδικημάτων. Τώρα για τη μελέτη αντικ... αντικτύπου φυσικά όλοι θέλουμε να, να έχουμε όσο το δυνατόν, να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα επιχειρήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω όμως ότι στη χώρα μου, όπως και σε άλλες χώρες, γνωρίζουμε πολύ καλά τι είναι η μελέτη των επιπτώσεων συχνά ε, οι μηνύσεις των γυναικών και οι καταγγελίες των γυναικών δεν λαμβάνονται σοβαρά στις χώρες μας. Ε, πολλές φορές οι δολοφονίες, οι ανθρωποκτονίες αυτές ε, είναι αναγγελθέντες εκ των προτέρων. δεν πρέπει λοιπόν να ασχολούμαστε μόνο για την ωραία διατύπωση στα νομικά μας κείμενα, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και την πραγματικότητα. Επομένως όλα τα επιχειρήματα είναι χρήσιμα, σίγουρα θα μας ε, πούν πολλά και οι συγητές και, σίγουρα επιδεικνύουν μια βούληση συνεργασίας την οποία εκτιμώ πάρα πολύ και ελπίζω ότι με τις τροπολογίες μου βελτιώνω το κείμενο και ελπίζω ότι η κυρία Χιμένες θα πραγματώσει αυτή τη φιλοδοξία να προστατεύσει όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα και να τους εξασφαλίσει αυτού του τύπου την προστασία. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αργήσει και να καθυστερήσει άλλο ένα τέτοιο ρυθμιστικό εργαλείο, γιατί στο κάτω-κάτω έχουμε κάνει πολλή δουλειά και σε άλλες κατηγορίες ατόμων που χρήζουν προστασίας. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δουλειά. Ευχαριστώ κυρία Κώστα. Δίνω το λόγο στην κυρία Γκρίσπετ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες και όλους τους συναδέλφους που έχουν ενδιαφερθεί εδώ και πολλές εβδομάδες για το θέμα αυτό που είναι τόσο πολύπλοκο. Εγώ θα είμαι σύντομη, συμφωνώ σε πολλά με την κυρία Κώστα και την κυρία Μπιλμπάου και νομίζω ότι είναι γνωστά όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να πείσουμε μεν τους δε ότι είναι απαραίτητο να καθοριστεί ένας τέτοιος χώρος προστασίας των θυμάτων στην Ευρώπη. Αυτό το ακούμε σε όλες τις συνεδριάσεις μας και τις συζητήσεις. Όλοι ομόφωνα συμφωνούμε να προστατευτούν τα θύματα. Είτε είναι γυναίκες, κυρίως γυναίκες είναι, αλλά θα ήθελα να προσθέσω όχι μόνο γυναίκες. Και με την έκθεση αυτή θα έπρεπε να καταλήξουμε στη δημιουργία ακριβώς αυτού του, αυτή μιας νομικής τάξεως προστασία. Δεν είμαστε όλοι πεπισμένοι, τόσο πεπισμένοι για το επίγον του θέματος βέβαια, γιατί ξεπερνάει τα, τις πολιτικάντικες διαφορές και έχει ενώ ξεπερνάει και έχει κάποιον επίγοντα χαρακτήρα από τη φύση του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη θέση ενισχύει της συνθήκης της Λισαβόνας καθιστά δεσμευτική νομικά τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μπορεί να θεωρούμε ορισμένοι ότι δεν έχουμε πλήρως καταλάβει το νόημά της, αλλά είναι βέβαιο ότι μας βοηθάει να προωθήσουμε αυτή την ιδέα της προστασίας των θυμάτων όπου και να βρίσκονται στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία καθώς και τον διπλό χαρακτήρα πρωτοτυπίας που έχει αυτή η εργασία γιατί πρώτον είναι κοινή με την Επιτροπή ΕΛΕΦ και δεύτερον νομική πρωτοτυπία που θύμισε η κυρία Κώστα ότι ζητούμε να ακολουθήσουμε ένα νομικό δρόμο που μας πρότειναν με τόλμη οι νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να υπάρξει δηλαδή καθαρά ενωσιακή δικαιοδοσία για την ιδέα αυτή και να προτείνουμε τη συγκεκριμένη προστασία των θυμάτων με ειδικό νομικό καθεστώς. Αυτό θα μας επέτρεπε να δείξουμε πόσο πρωτότυπες μπορούν να είναι οι ιδέες του Κοινοβουλίου με βάση πάντα αυτόν τον δεσμευτικό χαρακτήρα της χάρτας. Όπως είπε λοιπόν και η κυρία Πιλπάο, πιστεύω ότι είναι επίγον να ορίσουμε τώρα ένα χρονοδιάγραμμα, να σταματήσουμε να συζητούμε τις λεπτομέρειες, αλλά βασισμένοι στη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και όλοι μαζί, όλες μαζί να εφαρμόσουμε την ιδέα για την οποία συμφωνούμε, δηλαδή την προστασία των θυμάτων. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με το νομικό υπόβαθρο και οι προηγούμενοι και οι νομομαθείς αυτό μας είπαν. Μπορεί να είναι πρωτότυπη διαδικασία αλλά είναι σαφέστατη. Νομικά βέβαια στη συνέχεια είναι πολύπλοκη η εφαρμογή της και από τις τροπολογίες θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνουν εφαρμόσιμα όλα αυτά γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πλήρης σαφήνεια έτσι ώστε κάθε σε κάθε φάση της εφαρμογής της πρότασης η κάθε χώρα να μπορεί να λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα για να επιτρέπει την αποτελεσματικότερη προστασία των θυμάτων ή των δυνητικών θυμάτων αφού μιλούμε και για τους βουλγαρούς δημοσιογράφους ας πούμε ώστε τελικά να πάρουν όλα αυτά σάρκα και οστά όπως είπε και η κυρία Χιμένες στην εισαγωγή της, δηλαδή να υπάρξει αποτελεσματική προστασία τους και των μελλοντικών δυνητικών θυμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και τους συνα... τις και τους συναδέρφους για τις θέσεις τους. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην Ισπανική Προεδρία για να ακούσουμε τη θέση τους. Δίνω το λόγο στον κύριο Κολίνο κόμη; από την Ισπανική Προεδρία. Παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ συμπροεδρεύοντες. Στο παρελθόν, Είχα πει νομίζω ότι κάθε καινούριο πράγμα συναντά εμπόδια. Είναι ένα είδος ε, ψυχολογικού νόμου της ανθρωπότητας. Όλοι φοβούνται την αλλαγή, γιατί η αλλαγή σημαίνει αβεβαιότητα, αβέβαιο μέλλον και αυτό πάντοτε δημιουργεί εμπόδια. Είναι και ένας νόμος της φυσικής, είναι ο νόμος της αδράνειας, που σημαίνει αντίσταση στην απόπειρα κίνησης. Μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να, κάνει να κουνήσει κανείς τα, να ταρακουνήσει τα πνεύματα και να κινήσει την κατάσταση, να κουνήσει τα πράγματα. Και το συγκεκριμένο ζήτημα ε, είναι ακριβώς ένα τέτοιο παράδειγμα. Είναι η πρώτη φορά που ανταποκρινόμαστε νομοθετικά ε, σε κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Υπάρχει αυτή η αδράνεια, αυτή η αντίσταση στο να κουνηθούν τα πράγματα. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε ολοπλήρη στοιχεία και αριθμούς για τα ζητήματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία σε ορισμένα κράτη-μέλη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και μερικές άλλες χώρες, οι οποίες ε, αλλάζουν. Άλλες πάλι χώρες-μέλη δεν έχουν καθόλου τέτοιου τύπου στοιχεία. Εξαρτάται πώς ταξινομεί κανείς τα στατιστικά στοιχεία. Ε, σε ορισμένες χώρες ε, τα ε, εγκλήματα κατά των γυναικών δεν εντάσσεται στα έμφυλα δικήματα ή στα οικογενειακά δικήματα, αλλά στην ανθρωποκτονία και έτσι δεν γίνεται διαφοροποίηση και οι δύο εισηγητέ μας παρουσίασαν με πολύ ωραίο τρόπο το ζήτημα και το ανέφεραν το πρόβλημα αυτό με τα στατιστικά στοιχεία. Επίσης, τα νομικά προβλήματα δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα. Ε, έχουμε μία έκθεση από το Συμβουλίο και μία από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Το πρόβλημα δεν είναι η νομική βάση όμως. Ε, και οι δύο εκθέσεις, εάν και οι δύο εκθέσεις δεν συμφωνούσαν πάνω σε αυτό. Η Ισπανική Προεδρία δεν θα προωθούσε τα κείμενα αυτά. Έχουμε δύο λοιπόν γραπτά κείμενα από τη δική μας νομική υπηρεσία, από τη δική σας νομική υπηρεσία που είναι υπέρ της ε, σύνταξης μιας τέτοιας ε, έκθεσης, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει διαφωνία και διαμάχη για την νομική ε, βάση. Πόσες γνωμοδοτήσεις θα ζητήσουμε ακόμη από πόσες υπηρεσίες για να ξεκαθαριστεί αυτό. Έχουμε λοιπόν ήδη δύο κείμενα κείμενα, δύο νομοδοτήσεις που μας λένε ναι να προχωρήσουμε στην ε, έκδοση σχετικής νομοθεσίας, οπότε πρέπει να το κάνουμε. Και πράγματι ε, είναι και θέμα πολιτικής βούλησης. Υπάρχει πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό ή όχι. Υπάρχει πολιτική βούληση για να πούμε ότι οι εντολές προστασίας ε, που εκδίδονται σε μία εθνική επικράτεια θα πρέπει τώρα να ισχύουν σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Ναι ή όχι πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν είναι νομικό ζήτημα, αλλά είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και ποιο σώμα είναι πρόθυμο να ε, επιδείξει αυτή την πολιτική βούληση. Ε, όλα τα σχετικά ζητήματα πρέπει να διασαφινιστούν. Αλλά γι' αυτό ακριβώς γίνεται και αυτή η συζήτηση εδώ. Ήδη το είπαμε αυτό στην Προεδρία. Είμαστε σίγουροι ότι θα βελτιώσετε το κείμενο και γι' αυτό ακριβώς το συζητάμε. Σίγουρα το κείμενο του Κοινοβουλίου θα είναι πιο αποτελεσματικό, πιο σαφές και καλύτερο αν το καταφέρετε αυτό, είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε και να αποφύγουμε αυτή τη διπλή θυματοποίηση. Να μην γίνεται το ίδιο άτομο θύμα δύο φορές. Και σε ποια χώρα θα πρέπει να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, θα έλεγα σε όλες τις χώρες, ε, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν συμμετέχουν. Ε, υπάρχουν οι χώρες που δεν συμμετέχουν στο χώρο ελευθερίας και ε, δικαιοσύνης ίσως σε αυτό να θελήσουν να συμμετάσχουν και είναι φυσικά ελεύθερες να το κάνουν ή όχι. Οι άλλες χώρες όμως που αποτελούν μέλη του χώρου ελευθερίας και, και δικαιοσύνης θα πρέπει να το εφαρμόσουν. Ε, ε, κάτι άλλο θα ήταν παράλογο. Υπάρχουν ε, χώρες στις οποίες τρέχουν ποινικέ διαδικασίες για παράδειγμα, εντάξει θα ισχύει κάτι που ισχύει στην Ισπανία, θα ισχύει, θα ισχύει και στη Γαλλία, αλλά δεν θα ισχύει ίσως στην Αυστρία. Ε, υπάρχει αυτό το επιχείρημα ότι μπερδεύουμε την ποινική με την αστική δικαιοδοσία. Όχι, δεν ισχύει αυτό. οι αρχές πρέπει να κάνουν τα απαραίτητα. Πάντοτε το, το ίδιο ισχύει. Πρέπει να παρεμποδίζεται η διάπραξη εγκλημάτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ζήτημα λοιπόν ε, ποια αρχή είναι εκείνη η οποία θα κινεί τη διαδικασία, αν θα είναι οι ποινικέ αρχές ή αν θα είναι οι πολιτικές αρχές. Αυτό είναι κάτι που θα... Ε, ένα ζήτημα το οποίο θα επιληφθούν οι νομικές υπηρεσίες. Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα των διαφορετικών νομικών καταστάσεων και νομίζω, νομίζω ότι ήδη το κάνουμε. Δηλαδή αυτό το αργά ή γρήγορα είναι τώρα. Ε, κάποιοι μιλούν για βιωσιμότητα και για κατά πόσο θα διαρκέσει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι όταν μιλάει κανείς για ένομες καταστάσεις, όλοι μπορεί να έχουν την, τις αμφιβολίες τους. Υπάρχει το δικαίωμα στην αμφιβολία. Αλλά Υπάρχουν δύο εκθέσεις, δύο έγγραφα εδώ που μας λένε ότι δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε τουλάχιστον για τη νομική βάση. Τουλάχιστον αυτό. αν αμφισβητηθεί ακόμα και αυτό, τότε πρέπει να αναρωτηθούμε αν υπάρχει πολιτική βούληση. Εμείς στην Ισπανική Προεδρία, όπως θα θυμάστε, εμείς το επιφέραμε το ζήτημα στο προσκήνιο. Οπότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εμείς επιθυμούμε να προωθηθεί το ζήτημα. Έχουμε τώρα την πρόταση της Επιτροπής το 2011 ανάλογα από την φορά που θα πάρει η συζήτηση. Ε, ανάλογα, θα είναι μια ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, θα είναι κάτι που θα συμπεριλαμβάνει περισσότερα πράγματα. Αυτό θα απαιτήσει ακόμα περισσότερες συζητήσεις. Ε, δεν θα είναι, Δεν θα είναι εύκολη η υποδοχή μιας τέτοιας πρότασης. Θα υπάρχει αυτή η παρά επέκταση ή προστασία θυμάτων εκτός των συνόρων των κρατών μελών, εκτός της επικράτειας της ε, δικαστικής αρχής που εξέδωσε την νομική εντολή. Τώρα το άρθρο 3, 21 των συνθήκων. Υπάρχει μια προθεσμία, ε, τρεις μήνες νομίζω. Η ίδια προθεσμία για την προσχώρηση στον ε, ε, Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαίου, Ελευθερίας και Δικαιοσύνης. Τρεις μήνες. Το ίδιο είναι και με το άρθρο 21. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ρήτρα αποκλεισμού, έχει ρήτρα μη συμμετοχής. Ε, θα μας πούν βέβαια τι θα κάνουν οι Βρετανοί, θα επικαλιστούν αυτό το δικαίωμα μη συμμετοχή τους. Ε, θα πρέπει να μας το πούν μέσα σε τρεις μήνες, γιατί Μιλάμε 4 Ιουνίου που ήταν το Συμβούλιο μέχρι το Συμβούλιο του Οκτωβρίου που θα είναι η Βελγική Προεδρία. Θα πρέπει να μας πούνε λοιπόν αν θα συμμετέχουν ή όχι. Θα πρέπει αυτό να το δούμε στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Μόνο πέντε λεπτά έχω στη διάθεσή μου, οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να κρατήσω κι άλλο το λόγο. Ε, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, πλήρη εμπιστοσύνη στην πολιτική βούληση που έχει εκφραστεί μέσα από αυτή την κίνηση και έχω εμπιστοσύνη και στην Βελγική Προεδρία που θα ακολουθήσει πιστεύω ότι και εκείνη θα επιδείξει την ίδια πολιτική βούληση. Μετά από το ίμιση της Προεδρίας μας, στο επόμενο ίμιση της ε, Προεδρίας μας θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που είχαμε συμφωνήσει. Ευχαριστούμε τον κύριο Κόμπο από την Ισπανική Προεδρία για τις πληροφορίες αυτές από το Συμβούλιο. Και δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Φάου από την Κομισιόν για να ακούσουμε τις δικές του θέσεις. Παρακαλώ. Thank you, uh, Good Ευχαριστώ, Συμπρόεδρε. Καλησπέρα σας. Προφανώς το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Και δεν νομίζω, όπως είπε και η κυρία Μπιλμπά, ότι υπάρχει κανείς εδώ που να αμφισβητεί τη σημασία της χορήγησης βοήθειας βιώσιμης και μόνιμης ενός συστήματος προστασίας των θυμάτων ή δεχθών εγκλημάτων οπουδήποτε και να βρίσκονται. Συχνά βέβαια είναι νεαρά άτομα και ευάλωτα. Το μόνο θέμα είναι πώς να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα ρεαλιστικά η πολιτική θέληση είναι κάτι πολύ καλό, αλλά σε μια δημοκρατία ορίζεται από την ένομη τάξη. Και γι' αυτό, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, είναι σημαντικό ότι πρέπει να λειτουργήσουμε μέσα στα πλαίσια των συνθήκων. Δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε απλώς και μόνο γιατί θεωρούμε ότι κάτι είναι σωστό και μιλάω για όλα δηλαδή, τα ευρωπαϊκά όργανα, ιδιαίτερα όμως το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που είναι οι συνομοθέτε. Και η συνθήκη έχει κάνει μια, ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ ποινικού δικαίου και αστικού δικαίου. Έτσι είναι. Λοιπόν, έγιναν συζητήσεις σε πολλές χώρες μέλη πολλές φορές, πολύ, κατά την πολλές φορές δύσκολη διαδικασία έγκρισης της συνθήκης Λισαβόνας για να καθοριστούν ακριβώς οι δικαιοδοσίες της Ένωσης στο ποινικό δίκαιο το οποίο δεν ήταν εύκολο θέμα, ήταν, υπήρξε πολύ αμφιλεγόμενο. Πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε τις μάλλον αυστηρές διατάξεις ως προς αυτό των συνθήκων. Γι' αυτό το λόγο η πρόταση μιας ομάδας χωρών μελών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ποινικό δίκαιο της συνθήκης πρέπει να περιοριστεί μόνο στην καταπολέμηση ποινικών αδικημάτων και όχι και σε αστικά θέματα. Και δεν πρόκειται με την προσθήκη γενικών δηλώσεων των στόχων της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 3, αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Συγχωρείτε μα λοιπόν, αλλά εμείς διαφωνούμε με την νομική σας υπηρεσία. Λυπόμαστε γι' αυτό, αλλά νομίζουμε ότι δεν βασίζεται σε σωστή νομική πραγματογνωμοσύνη. Το Συμβούλιο απ' την άλλη θεωρεί ότι μόνο το άρθρο 88 χωρίς την προσθήκη του 3 της Λισαβόνας αρκεί και αυτό. Ούτε αυτό είναι σωστό. Εάν νομοθετούσαμε μόνο σε αυτή τη βάση θα δημιουργούσαμε κάτι που δεν επρόκειτο να εφαρμοστεί ποτέ. Με την πρώτη προσφυγή στα δικαστήρια θα καταστρεφόταν η νομοθεσία αυτή. Δεν πρόκειται για προστασία θυμάτων έτσι, αλλά απλώς για ένα βραχύβιο σύστημα που δεν δίνει στον κόσμο αυτό που χρειάζεται. Πολύ απλή απάντηση και αυτό απαντούμε στην έκκλησή σας, ώστε τα τρία όργανα να καταλήξουν σε ένα συμβιβασμό και σε συνένεση για να βρεθεί ο πιο ρεαλιστικός και βιώσιμος τρόπος υποβοήθησης των θυμάτων εγκλημάτων. Εσείς και το Συμβούλιο θέλετε να υπάρξει νομοθεσία για ποινικέ διαδικασίες ως καθεαυτές. Και να συμπληρωθεί αυτό μετά την προπαρασκευαστική εργασία το 11 ή όπως λέμε τώρα το 2011. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα χρειαστεί άλλη δέσμη μέτρων με διαφορετικό νομικό υπόβαθρο και διαφορετική σύνθεση της συμμετοχής των χωρών μελών στις διαδικασίες αυτές και θα έχει και πρόσθετο διοικητικό βάρος. Ξέρω ότι τα θύματα των εγκλημάτων δεν ενδιαφέρονται καθόλου να γνωρίσουν αυτά, αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά εμείς πρέπει να τις σεβαστούμε, γιατί έχουμε την ένωμη τάξη μας και δεν έχουμε ό,τι διαδικασία θέλουμε. Λειτουργούμε με τις συνθήκες. Συνθήκες που πρόσφατα είχαν τύχει τρομερών συζητήσεων. Αυτό θεωρεί λοιπόν η Κομισιόν ως τον ρεαλιστικότερο τρόπο. Αν θέλετε να περιοριστούμε μόνο στα αυστηρά ποινικά γίνεται από τώρα. Και στη συνέχεια μπορεί αυτό να συμπληρωθεί του χρόνου με πρόσθετη νομοθεσία για προστασία και άλλων τύπων αδικημάτων. Αλλά δεν γίνεται με μία ενιαία νομική βάση τόσο ευρεία είτε θα είναι υπερβολικά ευρύ ο στόχος για τη νομική βάση είτε το αντίθετο. Ίσως να είναι κρίμα αυτό, δεν γράψαμε εμείς τις συνθήκες, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Οι συνθήκες πρέπει να εφαρμοστούν και μάλιστα αυστηρά. Αλλιώς εμείς θεωρούμε ότι κάποιο δικαστήριο, ίσως και το ευρωπαϊκό, θα καταλήξει να κρίνει ότι η προτινόμενη νομοθεσία είναι αντισυνταγματική. Αυτό δεν θα ήταν καλό για κανέναν και η προστασία που θα θέλαμε να δημιουργήσουμε δεν θα ήταν ρεαλιστική ούτε σωστή. Ας κάνουμε τα πράγματα λοιπόν όπως πρέπει. Είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία των θεσμικών οργάνων θα βρει κάποιον τρόπο. Ίσως αυτό που σας λέω σε δύο φάσεις. Έτσι γίνεται, αυτά προβλέπει η συνθήκη. Όσο το δυνατόν συντομότερα βέβαια και όσο δυνατόν συνοπτικότερα για να είναι όλα ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα και να υπάρξει πραγματική προστασία των θυμάτων. Ευχαριστώ θερμά για τις απόψεις αυτές. Έχουμε ένα συνάδελφο ακόμα που ζήτησε το λόγο. Του δίνω λοιπόν το λόγο. Yo creo que el debate está bastante... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η συζήτηση έκλεισε και τώρα πρέπει να λάβουμε μία απόφαση. Δυστυχώς, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτού που θέλουμε εμείς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεδομένου αυτού που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχουμε άλλη επιλογή πρέπει να μην κάνουμε τίποτα και να περιμένουμε ε, να συντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα κείμενο σύμφωνα με μια σαφή νομική βάση που θα διακρίνει μεταξύ ποινικών και αστικών ζητημάτων. Αυτό είναι μία λύση. Μία λύση που σημαίνει, θα σημάνει το τέλος αυτών των εργασιών και την αναμονή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεύτερη επιλογή. Έχουμε δύο νομικές γνωμοδοτήσεις, μία του Κοινοβουλίου και μία του Συμβουλίου. Με αυτές τις γνωμοδοτήσεις ε, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Ας το κάνουμε λοιπόν. Ας πάρουμε μια απόφαση. Ε, αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να συζητούμε επί για το ζήτημα αυτό. Αυτές τις δύο λύσεις έχουμε. Και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο με την πρωτοβουλία του Συμβουλίου διαθέτει την απαραίτητη νομοθετική, το απαραίτητο νομοθετικό βάρος για να προχωρήσει. Ε, όπως έχει προτείνει το ΕΛΚ μπορούμε να υποβάλουμε και τις απαραίτητες τροπολογίες. Πολύ λογικό είναι. Μπορούμε να το συζητήσουμε με τις ε, κοινοβουλευτικές μας ομάδες, ο καθένας. Ε, κατανοώ ότι μπορεί στο πλαίσιο κάθε κοινοβουλευτική ομάδα ε, να υπάρχουν διαφωνίε κτλ. Αλλά το κάθε, κάθε κοινοβουλευτική ομάδα μπορεί να βάλει τάξη στο εσωτερικό τη, να το συζητήσει. Το Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλιστέ κτλ. Το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει. Δικαιούται να προχωρήσει. Ας το κάνουμε λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Εγώ αυτό προτείνω. Αν υπάρχει συμφωνία στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου για το κείμενο αυτό, ας το συντάξουμε και α θεωρεί η Επιτροπή ότι δεν πρέπει να το κάνουμε, εφόσον υπάρχει μια πολιτική βούληση, εφόσον έχουμε τις νομικές γνωμοδοτήσεις, εφόσον πιστεύουμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, ας το κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλει, ας, κάνει ό,τι θέλει και ας ολοκληρώσει τη δουλειά της στο επόμενο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά. Να δώσω το λόγο στις δύο εισηγήτριές μας. Πρώτα λοιπόν δίνω το λόγο στην κυρία Χιμένες. Παρακαλώ. Sí, eh, lo que quería decir que, bueno, otra vez repetir un poco lo que hemos dicho. Ναι, ίσως θα πρέπει να επαναλάβω αυτό που είπαμε όλοι. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Προσπαθούμε να διευκρινίσουμε κάποια ζητήματα, αλλά φαίνεται ότι βαδίζουμε με βήμα σημειωτών, ότι κάνουμε κύκλους. Όλοι θέλουμε η προστασία αυτή να προχωρήσει, αλλά δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι πρόκειται για πολιτική φύση θέμα. Συμφωνώ με όσους το πιστεύουν αυτό, διότι έχω συζητήσει με πολλούς στα θεσμικά όργανα, έχω συζητήσει με συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες και οι κίνδυνοι που υπάρχουν βρίσκονται ακριβώς στον πολιτικό χώρο. Μπορεί να υπάρχει φόβος ότι το μέσο αυτό δεν θα είναι αποτελεσματικό. Ο κόσμος δεν λέει ότι συμφωνώ με την Κομισιόν ή συμφωνώ με το Συμβούλιο. Ο κόσμος πιστεύει στην έκθεση αυτή, εγώ πιστεύω σε αυτήν και την στηρίζω με όλη μου την καρδιά. Αλλά όταν κάποιος μου λέει ότι αυτή θα οδηγήσει σε προβλήματα, Απορώ. Διότι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε αυτήν την εντολή προστασίας. Αλλά θα πρέπει επίσης να αναρωτηθούμε τι κάναμε λάθος και σκέφτομαι και εμένα εδώ, διότι εγώ έχω υποβάλει την έκθεση. Τι έχουμε κάνει λοιπόν λάθος και βρεθήκαμε στην παρούσα κατάσταση. Δεν πιστεύω ότι είναι πολιτικό θέμα. Δεν νομίζω ότι για πολιτικούς λόγους ο κόσμος ε, είναι αντίθετος με την πρόταση αυτή. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε υποστήριξη από όλες ε, τις ε, ομάδες. Αλλά τι κάναμε λάθος και βρισκόμαστε στην παρούσα κατάσταση. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτήν. διότι το οφείλουμε στα θύματα. Πώς προστατεύουμε τα θύματα της τρομοκρατίας, αλλά όχι ε, τις γυναίκες και τα παιδιά που μπορεί να γνωρίζουν και ε, τον δράστη. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσω. Εγώ ήθελα να Παρατείνω την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για να έχουμε μια όσο γίνεται πιο ευρεία έκθεση για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας, να μην χρειαστεί να την περιορίσουμε. Δεν θέλω να φρενάρω τις ε, διαδικασίες σε ένα θέμα ε, στο οποίο ήμουν υπέρ από την αρχή, αλλά υπάρχουν κράτη-μέλη που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να υιοθετήσουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας, διότι πιστεύουν ότι δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να ασκηθεί δίωξη κατά κάποιο δράστη. Έχουμε τις γνωμοδοτήσεις από τις νομικές υπηρεσίες, δύο γνωμοδοτήσεις, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι κατά του θέματος αυτού. Είναι ένα θέμα που πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας. Το όνομα μου θα βρίσκεται πάνω στην έκθεση αυτή και στο μέλλον θα βλέπω το θέμα αυτό, δεν είμαι ειδική στο θέμα αυτό. Φοβάμαι όμως ότι η έκθεση αυτή θα καταλήξει σε ένα σιρτάρι και δεν θα οδηγήσει πουθενά. Αυτό με ανησυχεί κυρίω. Πρώτη φορά θα έχω το όνομά μου πάνω σε μια έκθεση και θα ήθελα πολύ να είναι καλή η έκθεση αυτή και να οδηγήσει κάπου. Φαίνεται πως δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε εδώ πέρα, εγώ όμως ελπίζω ότι θα μπορέσουμε ελπίζω να μπορέσουμε να πετύχουμε και τη συμμετοχή της Κομισιόν, την υποστήριξη της Κομισιόν για την πρωτοβουλία αυτή. Όσον αφορά τις τροπολογίες, το είπα και αναφέρθηκε και εδώ, ότι η καλή ημερομηνία θα ήταν η 10η Ιουλίου. Θα ξεκινήσουμε πάλι τις εργασίες μας το Σεπτέμβριο. Θέλω να δω κάποια συνέχεια στο θέμα αυτό θέλω και κάποια χέγγια. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την Κομισιόν και δεν νομίζω ούτε ότι η Κομισιόν θέλει να μας αποσπάσει, να μας εμποδίσει να κάνουμε τη δουλειά μας. Νομίζω ότι όλοι ε, ε, ε, συμβάλλουν καλή την πίστη, αλλά πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Να δώσω το λόγο στην κυρία Ρομέρο για μια τελική παρέμβαση. Παρακαλώ. Señora Presidenta, cuando eh, la Comisión... Κυρία Πρόεδρε, η Κομισιόν ποτέ γραπτός βέβαια, ποτέ έκανε την πρότασή της για την οδηγία και πολλές φορές μας είπε ότι για να μπορέσει να εφαρμοστεί χρειάζεται κάποια απόφαση δικαστική και να έχει διαπιστωθεί το έγκλημα για να μπορέσει να χορηγηθεί βοήθεια. Ναι, αλλά αν έχει διαπιστωθεί το έγκλημα και έχει γίνει το έγκλημα δεν πρόκειται για πρόληψη πια. Εμείς μιλάμε για πρόληψη, δεν μιλάμε για τιμωρία, κύρωση. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε αρχίσει όλη αυτή τη διαδικασία προστασίας μελλοντικών θυμάτων. Η Κομισιόν Προσπαθεί εδώ να μας αποπροσανατολίσει. Αυτό κάνει. Αυτό μας αποπροσανατολίσει. Μια πρόληψη μιλάμε όταν λέμε προστασία. Βέβαια μπορούν οι χώρες να έχουν δικά τους μέτρα όπως γίνεται στην Ισπανία. Και όχι για ποινική μονοκύρωση. Τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν είναι πάρα πολλά. Επί 32 θεμάτων, θυμάτων στην Ισπανία μόνο 5 έχουν όμως υποβάλει μήνυση και εκ αυτών των 5 οι 4 την απέσυραν. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα πράγματα μόνο με τις κυρώσεις λοιπόν. Εδώ μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Για οικιακή και ιδιωτική τρομοκρατία. Και δεν είναι η πρώτη φορά που η τρομοκρατία πρέπει να αντιμετωπιστεί και με αστικό και με ποινικό τρόπο. Αν θέλουμε λοιπόν πραγματική προστασία των θυμάτων έναντι της ιδιωτικής τρομοκρατίας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί να, πάρ, να λάβουμε τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Εμένα η θέση μου είναι σαφής. Δεν πρέπει να αποσύρουμε την πρόταση αυτή, αλλά να επιμείνουμε. Και θα ζητήσω από όλες τις ομάδες να το σκεφτούν, να σκεφτούν δηλαδή πώς μπορούμε να προωθήσουμε το θέμα, να μην ξεχάσουμε όλα όσα κάναμε μέχρι τώρα και να έχουμε συνέστηση που έχουμε ήδη των ορίων που έχει η πρόταση αυτή. Και ένα μονοθήμα αν βοηθήσουμε καλό θα ήταν. Ευχαριστώ κυρία Ρομέρο. Πετύχαμε λοιπόν συμφωνία σχετικά με το εξής χρονοδιάγραμμα. 12 Ιουλίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. 2 Σεπτεμβρίου θα έχουμε τη συζήτηση για τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε 29-30 Σεπτεμβρίου. Μια προσανατολιστική ψηφοφορία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέρφους, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που συμπροεδρεύσαμε και να ευχαριστήσω και τη γραμματεία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για τη συνεργασία ανάμεσα στις δύο επιτροπές μας. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή Ισότητας θα συνεχίσει τη συνεδρίασή της. Please take Για καθίστε παρακαλώ. Λάβατε τα θέσεις σας, υπάρχουν θέσεις πίσω. Συνεχίζουμε λοιπόν τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας αν κοιτάξουμε την ημερησία διάταξη, βλέπουμε ότι το σημείο 2 είναι έγκριση της ημερησίας διάταξης. Δεν είχαμε αντιρρήσεις σε σχέση με το σχέδιο ημερησίας διάταξης. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερησία διάταξη. Σημείο 3. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Καταρχήν θα ήθελα στο όνομα της Επιτροπής να καλωσορίσω ανθρώπους της τοπικής διοίκησης από Ιταλικές περιφέρειες στην Πούλια, Καλαβρία και Αγιούσο που έχουν προσκληθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας από την κυρία Ματέρα. Σας ε, καλωσορίζω θερμά στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Επίσης θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη ότι στις 20-21 Ιουνίου εγκαινιάσαμε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας στο Βίλνιους. Είναι ένα θέμα που είχε απασχολήσει πολύ την Επιτροπή μας. Είχαμε εργαστεί με αφοσίες για το θέμα αυτό. Όπως τα γνωρίζετε, ε, η απόφαση έχει ληφθεί εδώ και πολύ καιρό σχετικά με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας. Έχουν ε, γίνει τα εγγένεια τώρα. Εγώ συμμετείχα στην συνάντηση στο Βίλνιους συμμετείχα στα επίσημα εγγένεια και μπορώ να σας ε, ενημερώσω ότι πέρα από τα επίσημα εγγένεια ε, είχαμε και κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, κάποιες συναυλίες και χθες το απόγευμα διάφοροι συμμετέχοντες μας ενημέρωσαν σχετικά με την κατάσταση στον τομέα της ισότητας. Ήταν αθρώα η προέλευση, ήταν πολύ καλή η διοργάνωση. Έγινε επίσης συνέντευξη τύπου με συμμετοχή πολλών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επίσης έγιναν ε, επιμέρους συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες. Η κυρία αυτή ήταν η ανακοίνωση της ε, Προέδρου. Η κυρία Τόμσεν κάτι έχει να προσθέσει. Παρακαλώ. Θα ήθελα... Θα ήθελα να συζητήσω τι έγινε το προηγούμενο μήνα στην Ολομέλεια που το ΕΛΚ πρότεινε να αποσύρουμε τις εκθέσεις της Ήλτα Φιγκερέιρο. Απογοητεύτηκα τόσο πολύ και εξεπλάγην και κατάλαβα ότι οι άντρες δεν παίρνουν τις γυναίκες στα σοβαρά, τις μεταχειρίζονται σαν παιδιά. Έξι χρόνια έχω εργαστεί στο κοινοβούλιο με ανθρώπους, με άντρες που έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις από μένα. Αλλά έμαθα ότι άσχετα από ε, που ανήκουν, είτε ανήκουν στο ΕΛΚ είτε στο ECR, ο λόγο ενό άντρα είναι λόγο ενό άντρα, αλλά τώρα φοβάμαι ότι με την έκθεσή μου στην Ολομέλεια θα μου φερθούν σαν παιδί. Ε, φοβάμαι ότι κάποιοι συνάδελφοι θα πούνε στην Ολομέλεια ότι δεν έχει τι απαραίτητε δεξιότητε. Ε, δεν ε, είσαι εξειδικευμένη και ότι η έκθεση αυτή που εκπώνησες βασίζεται σε εκθέσεις που ήδη έχουμε εκπονήσει, διότι η έκθεσή μου είναι γεμάτη από πράγματα που περιλαμβάνονται σε άλλες εκθέσεις. Φοβάμαι λοιπόν πολύ να βρεθώ στη θέση αυτή. και φοβάμαι πολύ σχετικά με τη φήμη της Επιτροπής Γυναικών, διότι ε, ούτως ή άλλως δεν μας πέρανε πολύ στα σοβαρά, τώρα πια σίγουρα καθόλου. Κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συζητήσουμε αν μπορούμε να έχουμε άλλες μεθόδους εργασίας, διότι δεν μου αρέσει καθόλου να γίνομαι ρεζίλη. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Τόμσεν. Η κυρία Μπάουερ επίσης ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Thank you so uh, Σας κατευχαριστώ. φαντάζομαι ότι θα το συζητήσουν και οι συντονιστές, αλλά αν μου δώσετε και μένα τη δυνατότητα να απαντήσω στην κυρία Τόμσον, θα ήθελα να απαντήσω. Θεωρώ ότι Το θέμα είναι κάπως ευρύτερο από το χρόνο που του διαθέσαμε. Είναι απογοητευτικό καμιά φορά να βλέπουμε, να συγκρίνουμε τι όντως συζητιέται στην Επιτροπή μας και τι λέγεται ότι συζητιέται. Καμιά φορά δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των δύο. Ποιο ήταν το κύριο θέμα, το κύριο θέμα λέγω. Ποιο ήταν ο λόγος για τον οποίο, για τον οποίο τα πράγματα έγιναν όπως έγιναν. Ο λόγος είναι ότι σε δύο εκθέσεις, δύο παράγραφοι ήταν ταυτόσιμες. Γιατί μάλλον προέρχονταν από την ίδια πηγή. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα ήταν τελείως απαραίτητο να προσέχουμε περισσότερο τι γράφουμε στις διάφορες εκθέσεις. Ε, είχα πει και πριν ότι δεν είναι σωστό σε κάθε έκθεση να τα βάζουμε όλα. Αυτό κάνουν πολλοί συνάδελφοι και συναδελφέ διότι έτσι καταρακώνουμε την αξιοπιστία της Επιτροπής μας. Γελιοποιούμαστε με αυτόν τον τρόπο, αν προσπαθούμε όλα να τα λύσουμε σε κάθε έκθεσή μας. Δεν είναι σωστός τρόπος αυτός. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να παραλείψουμε πολλά και έτσι να βελτιώσουμε τον τρόπο εργασιών μας. Καμιά φορά έχω το αίσθημα ότι μερικοί συνάδελφοι χρειάζονται περισσότερο πνεύμα συνεργασίας, περισσότερη πειθαρχία, καλύτερη εργασία συγγραφική των εκθέσεών τους, γιατί μερικές φορές εγκρίνουμε πολύ περίεργα πράγματα. μια από τις προηγούμενες εκθέσεις μας που σχεδόν αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα με αυτήν ζητούσε την εφαρμογή μιας νέας νομικής βάσης για κάποιο πρόβλημα ενώ ξέρουμε ότι καμιά φορά δημιουργούμε προβλήματα που δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν να, σας ευχαριστώ. Όχι, θέλω να προτείνω να επανέλθουμε και στους συντονιστές σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ. Ήθελα να σας προτείνω, επειδή αυτή είναι σημαντική συζήτηση, να την συνεχίσουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών την επόμενη φορά. Μία παρατήρηση ήθελα να κάνω. Όλα τα μέλη της Επιτροπής μας Έχουμε ευθύνη όχι μόνο να προωθούμε θέματα ισότητας, έχουμε και ευθύνη ώστε η Επιτροπή μας να ε, ενεργεί με τέτοιο τρόπο στο Κοινοβούλιο, ώστε να ενισχύουμε την ε, επιρροή μας στο Κοινοβούλιο. Κυρία Μπάουερ, ελπίζω να μπορέσουμε να επανέλθουμε στη συζήτηση αυτή στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών, διότι είναι πολύ σοβαρή. Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Το επόμενο θέμα είναι η έγκριση των πρακτικών των συνδριάσεων της 15ης Μαρτίου, της 16ης Μαρτίου και της 3ης και 4ης Μαΐου. Εάν δεν ακουστούν αντιρρήσεις ε, μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασής μας, θα θεωρηθεί ότι εγκρίθηκαν τα πρακτικά. Προχωράμε στο θέμα υπαριθμών 5 που έχει να κάνει με το ρόλο των γυναικών σε μια γυράσκουσα κοινωνία οι συντονιστές συμφώνησαν τον Σεπτέμβριο του 2009 να εκπονήσουμε την ε, έκθεση αυτή σύμφωνα με τον κανόνα 48. Πολύ θα ήθελα να ακούσω τις θέσεις της εισηγήτριάς μας, της κυρίας Πιέτη Κέινεν. Της δίνω λοιπόν το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω καταρχήν ότι το ζήτημα της γύρανσης γίνεται όλο και πιο ζωτικό στις κοινωνίες μας, γιατί η κοινωνία μας ολόκληρη γυράσκει, όπως ξέρουμε. Το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού στις ομάδες των ηλικιωμένων είναι γυναίκες. Επομένως είναι πολύ σε ένα γυναικείο ζήτημα. Δεύτερον, υπάρχει μια γενική στάση απέναντι στον όρο γύρανση. Συχνά το αντιμετωπίζουμε αρνητικά, ως ένα φορτίο ή ως ένα πρόβλημα είναι μια ετικέτα, μια ετικέτα που κάνει διακρίσεις εναντίον όλων των ηλικιωμένων μελών των κοινωνιών μας και αυτό ρίχνει μια μεγάλη σκιά στις υπηρεσίες μας αλλά και δεν αναγνωρίζει επαρκώς το γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι και οι συνταξιούχοι είναι σημαντικοί οικονομικοί παράγοντες, παρέχουν στην κοινωνία. παρέχουν με ανεπίσημους τρόπους στον ανεπίσημο τρίτο τομέα, στον τομέα παροχής βοήθειας. Πολλά μπορούν να γίνουν στα κράτη-μέλη και σε διάφορους θεσμούς για να δημιουργηθεί μια πιο θετική και δίκαιη στάση απέναντι στην ηλικία και στην αύξησή της. Επίσης, ένα άλλο γενικότερο ζήτημα είναι η τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση, η οποία έχει ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις ε, φυσικά για τον προϋπολογισμό και το δημόσιο χρέος των κρατών μελών. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες γενικά, οι ηλικιωμένοι και ιδιαίτερα οι ηλικιωμένες γυναίκες, ε, πολύ συχνά εξαρτώνται από τις ε, κοινωνικές υπηρεσίες και τα συστήματα προστασίας που εξαρτώνται από τον ε, προϋπολογισμό στις κοινωνίες μας. Επομένως, η οικονομική και κοινωνική κρίση πλήττει ισχυρότερα τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους, αλλά και ιδιαίτερα το πιο ευάλωτο τμήμα μεταξύ αυτών που είναι οι ηλικιωμένες γυναίκες. Και αυτό πρέπει να το, λάβουμε υπόψη μας και να λάβουμε και τα απαραίτητα μέτρα. Το τρίτο γενικό μου σχόλιο είναι ότι χρειαζόμαστε μια καλύτερη προσέγγιση ε, προς την γύρανση και προς τις ηλικιωμένες γυναίκες, όπως ακριβώς έχουμε μια σωστή βάση για την ισότητα των φύλων. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να δίνουμε ε, μια δεύτερη ή τρίτη άποψη για τη θέση των ηλικιωμένων. Αλλά οι ηλικιωμένοι και οι ηλικιωμένε γυναίκες συγκεκριμένα ε, έχουν ε, πρώτου βαθμού δικαιώματα στην κοινωνία μας και στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας και στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Συνταγματικών Δικαίων πρέπει να βλέπουμε τους ηλικιωμένους και τις ηλικιωμένες γυναίκες ως φορείς δικαιωμάτων, ως υποκείμενα δικαιωμάτων πρώτου βαθμού. Θα πρέπει λοιπόν η οδηγία κατά των διακρίσεων να τροποποιηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα και να χρησιμοποιηθεί ως ε, ένα ισχυρό εργαλείο για την διασφάλιση των συνταγματικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών μας. Συχνά οι διακρίσεις αυτές, οι οποίες μπορεί να έχουν πολλές πτυχές, είναι, είναι πολύ λεπτές διακρίσεις. Ε, ε, συνήθως ε, ο κόσμος αλλά και οι υπηρεσίες δεν συνειδητοποιούν ότι αρνούνται υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους δεν συνειδητοποιούν τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών. Χρειάζεται μεγαλύτερη έρευνα και ένας μηχανισμός παρακολούθησης των διακρίσεων κατά των ηλικιωμένων και των διακρίσεων κατά συγκεκριμένου φύλου. Πρέπει, πιστεύω, να εγκαθιδρυθεί μια τακτική μέθοδος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να ακολουθήσει και το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Πρέπει να υπάρξει μία μέθοδος όπου οι διακρίσεις κατά των ηλικιωμένων και οι διακρίσεις κατά συγκεκριμένου φύλου θα παρακολουθούνται και θα καταγράφονται και θα πρέπει να καταγράφεται ο τρόπος που ενεργούν οι κυβερνήσεις αλλά και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταγράφονται όλες εκείνες οι περιπτώσεις όπου αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν με το σωστό τρόπο αυτά τα τμήματα του πληθυσμού. Ε, υπάρχει και το θέμα των γυναικών με ειδικέ ανάγκες, αλλά δεν θα επισέλθω τώρα σε αυτό. Υπάρχουν οι πιο ηλικιωμένες γυναίκες ε, στον εργοσιακό βίο. Υπάρχουν οι διακρίσεις ε, στο χώρο εργασίας. Ε, τυπικά απαγορεύονται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν, γίνονται τέτοιες διακράσεις. Υπάρχει αυτό το γυάλινο ταβάνι. Είναι δύσκολο για τις πιο ηλικιωμένε γυναίκες, για τις μεγαλύτερες γυναίκες ε, να αναρριχηθούν στην ιεραρχία σε σχέση με τους ε, άντρες συναδέλφους τους και επιπλέον όταν ε, υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των γυναικών άνω των 40 ή των 50 ετών. Είναι πολύ πιο δύσκολο για αυτές να βρουν δουλειά σε σύγκριση με τους συνομιλίκους άντρες. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί και πρέπει να υπάρξει και μια σωστή παρακολούθηση και θα πρέπει να ληφθούν και μέτρα. Δύο άλλα σημεία. Υπάρχει η σύνταξη, η συνταξιοδότηση. Η σημερινή γενεά, νέα γενιά ονομάζεται σωτήρας. Ε, δουλεύουν λιγότερο γιατί φροντίζουν τα παιδιά τους και συχνά φροντίζουν και τους ηλικιωμένους ε, γονείς ή συγγενείς τους. Η, η σύνταξή τους όμως παραμένει χαμηλή. Χρειάζεται μια καλύτερη προσέγγιση στο σύστημα συνταξιοδότησης. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο το γενικό κόστος των συντάξεων στην κοινωνία μας, όπως συχνά συνηθίζεται σήμερα, αλλά πρέπει να δούμε και πώς, ε, τι αποχρώσεις υπάρχουν. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις διάφορες αποχρώσεις. Μακροπρόθεσμα θα ήταν καλύτερο αν τα κράτη-μέλη μπορούσαν να λάβουν κάποια μέτρα όπως είναι η γονεϊκή άδεια. Νομίζω ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να υπάρχει μια τέτοια προσέγγιση. Then, um, when it comes to next uh, uh, Λοιπόν, αν μιλήσουμε τώρα για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, σκέφτομαι τις υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Και εκεί, όταν προγραμματίζονται και οργανώνονται οι υπηρεσίες αυτές, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προσπελασιμότητα σε αυτές. πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα αυτών των ομάδων του πληθυσμού που φροντίζουν τους άλλους ε, να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στο σπίτι τους. Θα πρέπει επίσης το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των ε, παθήσεων της τρίτης ηλικίας ε, να προχωρήσει περισσότερο στην εφαρμογή του. Όταν δούμε τα συστήματα υγείας θα δούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα για τις ε, συμβουλές ως προς τη διατροφή και τις ιατρικές συμβουλές. Πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε ότι τα συμπτώματα των καρδιοναπνευστικών παθήσεων είναι διαφορετικά ε, στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες. Επίσης, ο καρκίνος του ορθού και του παχαίου σεντέρου μπορεί να έχει διαφορετικά συμπτώματα στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες. Τα αναφέρω ως παράδειγμα. Τις αναφέρω ως παράδειγμα αυτές τις νόσους. Επίσης, χρειαζόμαστε και πόρους τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κράτους μέλους για να επιταχύνουμε τις καινοτομίες που μπορούν να αποβούν σε όφελος. Για παράδειγμα, έχουμε τις τεχνολογίες, έχουμε την ψηφιακή ατζέντα. Μπορούν και αυτά τα εργαλεία να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους και τις ηλικιωμένες γυναίκες ειδικότερα. Και αυτό σε συνεργασία με τους χρήστες, μαζί τους, να κάνουμε κάτι μαζί τους και όχι για εκείνους. Καλό θα ήταν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα σχέδιο δράσης μέχρι το τέλος του έτους για, την, για τους τους πόρους που θα μπορούσαμε να διαθέσουμε για την ε, επιστημονική παρακολούθηση της τρίτης ηλικίας, για την αύξηση της ε, συνοχής και της συνάφειας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, της συντάξης, ε, να υπάρξουν διευθετήσεις μερικής απασχόλησης, να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα των μελών της τρίτης ηλικίας, να μην υπάρχουν διακρίσεις να υπάρξουν και άλλα μέτρα, όχι μόνο νομοθετική φύσεως για τη συνειδητοποίηση των αναγκών των ηλικιωμένων, όπως ενημερωτικές καμπάνιες κτλ. Άκουσα πολύ προσεκτικά ε, τη συνάδελφο, την κυρία Μπάουερ, για την οποία τρέφω το μεγαλύτερο σεβασμό. Ε, νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί εδώ και μια ευρωπαϊκή οδικία για τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες ε, προς όφελος των συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων. Υπάρχουν και άλλα θέματα που θα μπορούσα να θίξω, αλλά θα ήθελα να σταματήσω τώρα και να υπάρξει χρόνος για ερωτήσεις και παρεμβάσεις από τους συναδέλφους. Είμαι πολύ ανοιχτή ε, για να δεχθώ όσο το δυνατόν περισσότερα σχόλια και ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ την εισηγήτρια, την κυρία Κέινεν, για τις θέσεις αυτές. Στον κατάλογο των ομιλητών έχω πρώτα την κυρία Κορνέλισεν και κατόπιν την κυρία Τόμσεν. Παρακαλώ, πρώτα η κυρία Κορνέλισεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Βρίσκω πολύ καλή την έκθεσή της. Είδα μια προηγούμενη εκδοχή της που αντιμετωπίζει τα που ασχολείται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ε, ηλικιωμένε γυναίκε, οι γυράσκουσε γυναίκε στην κοινωνία. Η νέα βερσιόν όμω συμπεριλαμβάνει και κάποια προβλήματα αλλά και τι ευκαιρίε που ε, σε γυράσκουσες γυναίκες η δημογραφική αλλαγή. Θα ήθελα να πω ότι η δημογραφική αλλαγή είναι, αποτελεί γεγονός και ξέρουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε περισσότερους ηλικιωμένους και λιγότερους νέους. Αυτό δεν θα είναι αυτό καθ' αυτό πρόβλημα, εάν προβλέψουμε αρκετά την κατάσταση και προετοιμαστούμε για αυτήν. Τέλος, θα είναι χρήσιμο να εξετάσουμε τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν οι γυράσκουσες γυναίκες, διότι η ομάδα αυτή μεγαλώνει. Ε, ιδιαίτερα με ενδιαφέρει ε, η καταπολέμηση της διάκρισης για λόγους ηλικίας. Νομίζω ότι αυτός είναι ξεχασμένος λόγος διακρίσεων. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οι απαιτήσει ως προς την υγεία, προσοχή που δίνεται, δεν δίνεται αρκετή προσοχή στις γυναίκες ε, στην έρευνα στον τομέα της υγείας. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ε, στα νοσήματα που αναφέρθηκαν ε, την αρθρίτιδα, διότι πιο πολλές γυναίκες υποφέρουν ότι υπάρχει την ασθένεια αυτή από ότι άντρες δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα ασθένεια, πολύ λίγα χρήματα δίδονται για την έρευνα και δεν ε, είναι εμφανής η θέση στις στα ερευνητικά προγράμματα. Η φτώχεια φυσικά είναι πρόβλημα. Αλλά επίσης μας ενδιαφέρει να δοθεί προσοχή ε, στην θελοντική εργασία των ηλικιωμένων γυναικών ε, που αποτελεί μέρος της συμβολής τους, της συνεισφοράς τους στην κοινωνία. Επίσης, μου αρέσει το γεγονός ότι αναφέρεται το βάρος που φέρνουν οι γυναίκες ε, που ε, ε, εργάζονται. Θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Βρίσκω λοιπόν ότι το σχέδιο δράσης είναι εξαιρετική η ιδέα να το επιδιώξουμε και ελπίζω η Κομισιόν να το ολοκληρώσει. Είναι κάτι που στηρίζομαι όλοι με την καρδιά. Μια ερώτηση έχω, διότι βρίσκω ότι είναι σημαντική η έκθεση αυτή και θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή της Επιτροπής Απασχόλησης και Περιβάλλοντος στο θέμα αυτό. Έχει ζητηθεί η γνωμοδότησή τους ε, ή θα μπορέσουν να συμμετάσχουν με κάποιο άλλο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κορνέλισεν. Παρακαλώ κυρία Τόμσεν. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί τόνισε ιδιαίτερα αυτό το σημαντικότατο θέμα για τις ηλικιωμένε οι οποίες είναι και αυτές αθέατες, αόρατες από την κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να τις τονίσουμε, να τονίσουμε την κατάστασή τους περισσότερο, διότι γενικά οι ηλικιωμένοι είναι τομέας όπου δικαιολογείται να μιλάει κανείς για, την φιλογενε... για τη διάσταση των φύλων. Γιατί τα προβλήματα των γυναικών στην τρίτη ηλικία είναι διαφορετικά από των αντρών. Η δημογραφία έχει αλλάξει πολύ. Σήμερα υπάρχουν πολύ περισσότερες ηλικιωμένες από ό,τι ηλικιωμένοι και το 2025 10% του πληθυσμού της Ευρώπης θα είναι πάνω από 85 ετών. Και από αυτό το 10% 90% θα είναι γυναίκες. Το 9% δηλαδή. Και μάλιστα πτωχές. Διότι η σχέση τους με την αγορά εργασίας είναι άλλοι από τον αντρών γιατί είτε εργάζονται μερικώς είτε είναι μητέρες και οικοκυρές και γι' αυτό έχουν πολύ λίγες συντάξει και χρήματα και έσοδα. Και πολλές από αυτές τις γυναίκες εξαρτώνται από το δημόσιο για την ζωή τους για την επιβίωσή τους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα, μια πολιτική στην ένεση για τους ηλικιωμένους και να τους προσέξουμε ιδιαίτερα, ιδιαίτατα όμως τις γυναίκες που θα αποτελέσουν τεράστιο πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ κυρία Τόμσεν. Να δώσω το λόγο στην κυρία Παλιαδέλη, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης στην έκθεση αυτή και ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια που την ολοκλήρωσε ακόμη και σε αυτή την προκαταρκτική της μορφή. Είναι μεγάλο θέμα η γύρανση των κοινωνιών και των ανθρώπων στις γυράσκουσες κοινωνίες Ιδιαίτερα δε οι γυράσκουσες γυναίκες, της γυράσκουσες κοινωνίες των γυρασκών των ανθρώπων. Στο, σε, σε κοντινό μέλλον θα αυξηθούν οι αριθμοί των ηλικιωμένων. Γι' αυτό νομίζω ότι η πρότασή σας να γίνει μια επιστημονική έρευνα για την γύρανση του πληθυσμού και τις επιπτώσεις της, όχι μόνο δημοσιονομικά και οικονομικά, αλλά κυρίως τις υπόλοιπες κοινωνικές και ψυχολογικές πτυχές είναι πολύ καλή. Θα ήθελα να σχολιάσω τώρα τον τίτλο της έκθεσης. Τι λέει ακριβώς. Ο ρόλος των γυναικών σε μια γυράσκουσα κοινωνία όπως λέτε είναι η πραγματικότητα ή ο ρόλος των ηλικιωμένων γυναικών στη γυράσκουσα κοινωνία. Ίσως είναι καλύτερος αυτός ο δικός μου ο τίτλος. Από νομικής απόψεως τα σημεία 21 και 25 της συνθήκης της Λισαβόνας δικαιολογούν την ύπαρξη της έκθεσης αυτής. Έχουμε το δικαίωμα να ασχοληθούμε και είναι σημαντικό να δούμε κατά πόσον μπορούν ρεαλιστικά να εφαρμοστούν τα άρθρα, τα σημεία αυτά. στις διάφορες ευρωπαϊκές μας κοινωνίες που έχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμη μια έρευνα και η καθορισμός ορισμένων πυροτύπων ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να προσαρμόσουν τα συστήματά τους προς μια πιο ρεαλιστική και συντονισμένη με ένα πιο ρεαλιστικό και συντονισμένο τρόπο. Έχουμε δει πολλές φορές ότι υπάρχουν τέτοιες διαφορές στις κοινωνίες μας και πρόσφατα η οικονομική κρίση και η καθυστερημένη έκφραση αλληλεγγύης σε επίπεδο Κομισιόν, όχι Κοινοβουλίου, έδειξε ότι ακόμη πολλά μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν για να αυξηθεί η ευαισθησία μας, η ευαισθησία μας τα κοινωνικά όπως τη γύρανση των γυναικών σε ένα, μια γυράσκουσα κοινωνία. Είναι κρίμα αλλά ισχύει ότι οι ηλικιωμένοι όπως είπατε συνήθως θεωρούνται ως παθητικά αντικείμενα και όχι ως ενεργητικά υποκείμενα. Εκτός από όταν τους βλέπουμε ως καταναλωτές και καταναλώτριες. Τότε ναι, τότε ναι. Αλλιώς θεωρούνται απλώς παθητικά αντικείμενα. Από αυτή την άποψη λοιπόν τα γυροκομεία και το προσωπικό τους δεν πρέπει απλώς να επιμορφώνονται όπως είπατε αλλά και να επιμορφώνονται στην μεταχείριση των ηλικιωμένων. Έχω δει ανθρώπους να γυράσκουν πολύ γρηγορότερα αν δεν τους χορηγείται καμία συμμετοχή σε εκδηλώσεις, σε προετοιμασία του φαγητού των κλπ. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε και τον τρόπο με τον οποίο θεωρούμε τη λειτουργία ενός γυροκομείου, όχι ως απλό ίδρυμα που υποκαθιστά το νοσοκομείο, αλλά ως ένα χώρο όπου οι ηλικιωμένοι να μπορούν να διασκεδάσουν τη ζωή τους και να τη διαχειριστούν περισσότερο. Επίσης συμφωνώ απόλυτα με την εισηγήτρια ότι χαμηλότερες συντάξεις συνήθως προκύπτουν από το ότι οι γυναίκες έχουν χαμηλότερους μισθούς γενικότερα. Ιδιαίτερα διότι όπως λέτε η περίθαλψη που τους χορηγείται για τα παιδιά πάβει να υπάρχει όταν γεράσουν. Οι περισσότεροι υπάρχει όσο εργάζονται και όχι όταν γεράσουν. γιατί στην ενεργό ζωή τους έχουν ασχοληθεί και με τους γονείς τους και με τα παιδιά, είναι πάντοτε μεταξύ δύο γενεών οι γυναίκες. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη συνταξιοδότηση. Από αυτή την άποψη λοιπόν θα ήθελα στην τελική της μορφή η έκθεση αυτή να κάνει μία πιο τολμηρή σύσταση για ορισμένες κοινωνίες, όχι όλες για ορισμένες, για καλύτερη μεταχείριση αυτών των γυναικών που προσπαθούν να αναλάβουν όσο καλύτερα γίνεται αυτόν τον δύσκολο ρόλο που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες. Αυτές τις σύντομες σκέψεις θα τις συμπληρώσω τώρα παραδεχόμενοι ότι όντως οι ηλικιωμένες γυναίκες συμβάλλουν στην, στον κοινωνικό τους περίγυρο και δεν πρέπει αυτό να μείνει χωρίς κάποιο είδους αποζημίωση. Πρέπει να υπάρξει κάποιος τρόπος η συμβολή των γιαγιάδων με ή χωρίς εισαγωγικά, δηλαδή ηλικιωμένων γυναικών που είναι διατεθειμένες να παίξουν το ρόλο της γιαγιάς φροντίζοντας παιδιά, νομίζω ότι θα ήταν κάτι πολύ θετικό για την κοινωνία γενικότερα. Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι οι γιαγιάδες. για την ασφαλή ανατροφή των παιδιών. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις ηλικιωμένε γυναίκες με τρόπο που να στηρίζει την κοινωνία και την οικογένεια και τις εργαζόμενες γυναίκες που θα βοηθούνταν έτσι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καριέρας τους με πιο ελεύθερο τρόπο αν ήταν σίγουρες ότι γυρεότερες γυναίκες θα είναι παρούσες για να χορηγήσουν στα παιδιά την τρυφερότητα που τους χρειάζεται όταν λείπουν οι μητέρες των. Αυτά όλα πρέπει να πληρώνονται κάπως. Κάπου λέει εδώ στο 3 νομίζω. Το 3 νομίζω πρέπει όμως να το λέει πολύ πιο δραστικά ότι το 12 πρέπει να εορταστεί ως έτος ενεργούς γυράνσεως. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό σημείο της έκθεσης και συγχαίρω την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Μπάουερ. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα γενικότερου ενδιαφέροντος και ότι έχει έρθει η ώρα να στρέψουμε την προσοχή μας πάνω σε αυτό. κάποια σχόλια ή ερωτήσεις για την έκθεση αυτή. Στο άρθρο 5. Νομίζω ότι εκτός από τα μέτρα που προετοιμάζονται κατά των διακρίσεων, Έχουμε αρκετές τέτοιες οδηγίες, τουλάχιστον δύο. Μία για, την εργασιακή, για εργασιακό βίο και μία για την πρόσβαση στις υπηρεσίες και στην απασχόληση. Νομίζω ότι δεν έχουμε αρκετή γνώση, δεν έχουμε αρκετές γνώσεις για το πώς λειτουργούν στην πράξη αυτές οι οδηγίες. Έχω την αίσθηση, αλλά δεν το έχω ελέγξει, έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή το Ίδρυμα του Δουβλίνου ήρθε σε επαφή πριν από μερικά χρόνια, ε, εν πάση περιπτώσει όχι πριν από πολύ καιρό, ίσως πριν από ένα με δύο χρόνια, ήρθε σε επαφή με κάποιους ερευνητές, ε, με κάποια έρευνα για τις διακρίσεις κατά των γυναικών ή τέλο πάντων ε, αυτό ως τμήμα άλλων ερευνών για την αγορά εργασίας τη διασύνδεση της αγοράς εργασίας και την ηλικία. Θα ήταν χρήσιμο να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εμείς. Όπως και να έχει, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη προσοχή τη λιγότερη ασημένια οικονομία. Ε, ε, Πρέπει να δούμε λίγο αυτήν την ε, μερίδα των γυναικών που είναι αποφασιστική, όχι μόνο από πλευράς κατανάλωσης, αλλά και από πλευράς παροχέων υπηρεσιών. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Και εκτιμώ το γεγονός ότι σύμφωνα με την εισηγήτρια κάτι τέτοιο θα προσέφερε έντονη προστιθέμενη αξία. Ίσως θα έπρεπε να ζητήσουμε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από τον Οργανισμό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να ζητήσουμε κάποιες, μια έκθεση ή να ζητήσουμε να ενημερωθούμε για τις εκθέσεις ε, σχετικά με τις διακρίσεις κατά των ε, ηλικιωμένων. Νομίζω ότι είναι περισσότερο δική του αρμοδιότητα παρά αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω μία ερώτηση και για το άρθρο 24. Δεν ξέρω αν ε, η μετάφραση είναι καλή. Ε, μερικές φορές έχουμε προβλήματα με τις μεταφράσεις. Πώς πρέπει κανεί... Ε, υπάρχει αυτή η φράση για την εγγύηση του βασικού εισοδήματος. Από όσο ξέρω η κυρία Φιγερέιδο είναι στην Επιτροπή Απασχόλησης και έχει μια έκθεση για το ελάχιστο εισόδημα. Νομίζω ότι είναι προβληματικό αυτό. Τι θα πει να εγγυηθούμε το δικαίωμα στο κατώτατο εισόδημα. Ίσως πρέπει να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ, η κυρία Μωρίν. Merci, Madame la Présidente. Je crois que... Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί πράγματι γιατί ουσιαστικά έχει να κάνει με τη γύρινση του ευρωπαϊκού πληθυσμού από τη μία πλευρά, αλλά και με την παράταση της ζωής ε, που αφορά πολύ περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άντρε, γιατί ξέρουμε ότι σήμερα ένα από τα δύο κοριτσάκια που γεννιούνται θα ζήσει πάνω από 100 χρόνια. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ ειδικό πρόβλημα μπροστά μας, ειδικό όχι μόνο της ευρωπαϊκής κοινωνίας, αλλά ειδικό για τις γυναίκες μέσα στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Θέλω να επανέλθω βέβαια ακόμα και στον τίτλο της έκθεσης. Ο ρόλος των γυναικών στο πλαίσιο ενός γυράσκοντος πληθυσμού. Ο ρόλος των γυναικών λοιπόν. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό το λέει η έκθεση στην αρχή της. Μιλά για, την, για τις νοοτροπίες απέναντι στην γύρανση. Όπως το είπε και η κυρία Μπάουερ στην αρχή, μια κοινωνία που γυράσκει δεν είναι μια κοινωνία παραμερισμένη, αλλά σήμερα με, την, με το προσδόκιμο μιας ακόμα, ενός ακόμα μεγαλύτερου βίου ε, θα είναι μια ομάδα που θα εξακολουθεί να δραστηριοποιείται περισσότερο. Πρέπει λοιπόν όχι μόνο να αλλάξουν οι νοοτροπίες, αλλά να βρεθούν και καινούργοι τρόποι ένταξης, συμπερίληψης αυτού του γυράσκοντος πληθυσμού για να μην αφαιθεί ο πληθυσμός αυτός έξω από τον ενεργό βίο. Το δεύτερο σημείο πάνω στο οποίο θα είμαι πολύ σύντομη γιατί πολλά υπόθηκαν ήδη. Το δεύτερο λοιπόν σημείο που ήθελα να θίξω αφορά ένα ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο έχει διατυπωθεί το σημείο 11. Στο σημείο 11 ε, ζητούμε η γυναίκα να αυξηθεί ο αριθμός αμοιβόμενης εβδομαδιαίας απασχόλησης για τις γυναίκες. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάτι πολύ το θετικό σε αυτό, αλλά θα ήθελα να τα πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Οι γυναίκες στην ουσία σε όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου για πολλούς και διάφορους λόγους ειστερούν χρονικά σημαντικά στις μισθολογικές τους αποδοχές και όταν φτάνουν στην ηλικία της συνταξιοδότησης ή στο τέλος του επαγγελματικού τους βίου ε, εμφανίζονται απαράδεκτες μισθολογικές αποκλίσεις. Πρέπει λοιπόν να αγρυπνήσουμε, να είμαστε σε εγρήγορση για τον τρόπο που θα διατυπώσουμε αυτή την παράγραφο. Δεν πρέπει να, να μας δώνει να καταλάβουμε το αντίθετο από αυτό που επιδιώκει. Πρέπει πολύ μεγάλη προσοχή να δώσουμε στην ε, διατύπωση μιλάει για μισθολογική απόκληση 30%. Σίγουρα υπάρχουν σημαντικές μισθολογικές αποκλήσεις και αυτές πρέπει να αντιμετωπισθούν με άλλο τρόπο και όχι μόνο με αύξηση του χρόνου εργασίας. Διαφορετικά, εμείς είμαστε οι πρώτες που θα δεχτούμε ότι πρέπει να εργάζονται περισσότερο. Είμαστε οι πρώτες που θα πούμε ότι οι γυναίκες στην ουσία δουλεύουν περισσότερο από τους άντρες. Για να κερδίσει μια γυναίκα σήμερα τον ίδιο ε, μισθό ε, μέσα σε ένα έτος, η γυναίκα πρέπει να δουλέψει πολύ περισσότερο. Πρέπει να δουλέψει και κομμάτι του επόμενου έτους για να έχει επιτύχει τον ίδιο μισθό. Αν λοιπόν η συγγήτρια θέλει να καταγράψει αυτό το σχόλιο, Ζητούμε επίσης την προαγωγή πιο ευέλικτων χρόνων εργασίας, επίσης μεγαλύτερα, περισσότερα συμβόλαια ε, περιορισμένης απασχόλησης. Ε, κατ' εμέ το σημείο αυτό, το σχόλιο αυτό, ε, δεν βρίσκεται στο σωστό σημείο. Εγώ προσωπικά θα το έβαζα στο σημείο 12. Γιατί? Γιατί βλέπουμε πολύ καλά ότι σε μια γυράσκουσα κοινωνία πρέπει να επινοήσουμε νέα μοντέλα άδειας ε, για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία ε, για τους υπεύθυνους παροχής φροντίδας τους ηλικιωμένου. χωρίς όμως να συσσωρεύονται και πάλι καθυστερήσεις στον επαγγελματικό βίο ε, και στις μισθολογικές απολαβές. Νομίζω λοιπόν ότι εγώ συμφωνώ με τις νέες αυτές μορφές άδειας, γιατί σήμερα σε πολλές χώρες οι γυναίκες έχουν δικαίωμα άδειας για να, να ασχοληθούν με τα παιδιά τους, αλλά δεν έχουν δικαίωμα άδειας για να ασχοληθούν με άτομα της προηγούμενης γενιάς. Και αν τους δοθούν τέτοιες άδειες, πολύ φοβάμαι ότι θα συσσωρευθούν νέες καθυστερήσεις. Γι' αυτό και ζητώ, γι' αυτό θα ήθελα οι νέες μορφές άδειας και τα οι ευέλικτες μορφές εργασίας να συμπεριληφθούν σε αυτήν την έκθεση αλλά σε άλλο σημείο. Να είμαστε πολύ προσεκτικές λοιπόν. Έχουμε μια πραγματική ευθύνη εδώ. Μερικές φορές, ξέρετε, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Πρέπει να προσέξουμε ε, να μην να μην τελικά στραφούμε κατά των γυναικών στις πολυθεμητές μας επιδιώξεις. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Οβίρ. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ ήθελα να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο σημείο, το σημείο 24. Η κυρία Πάουερ όμως ήδη το ανέφερε, γι' αυτό δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω. Ωστόσο, δεν είναι σαφές τι είναι ε, το εγκυμένο εισόδημα με βάση το βασικό εισόδημα που θα εξαρτάται από το επίπεδο ζωής του κράτους μέλους. Ίσως ε, θα μπορούσαμε να μιλάμε για έναν ελάχιστο μισθό, ο οποίος διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Βέβαια καταλαβαίνω όμως ότι όλοι ε, γυράσκουμε, δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από αυτό και η διαφορά στις ε, απολαυές ανδρών και γυναικών έχει αυξηθεί. Ε, Ήταν 14% πριν κάποια χρόνια, τώρα είναι 17%. Ε, περνάμε οικονομική κρίση, τι θα γίνει μετά από αυτήν δεν το γνωρίζουμε. Ε, αλλά θα επηρεαστούν οι συντάξεις. Θα συζητήσουμε άλλη έκθεση για την ε, γονική άδεια. Δεν έχω ακούσει ακόμα κανέναν να ρωτάει Γιατί μια γυναίκα που παίρνει γονική άδεια δεν παίρνει το 100% του μισθού της κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας. Ξέρετε, οι γυναίκε παίρνουν μικρότερες συντάξεις από τους άντρες, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα κάποιων συγκυριών. Θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι γι' αυτό και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες στα έγγραφά μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι ολοκληρωμένη, πλήρης, ε, διότι δεν περιγράφει μόνο την κατάσταση, προτείνει και λύσεις. Είμαι συνεισηγήτρια της ΑΛΤΕ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους... Θα ήθελα να ακούσω και τους άλλους συνεισηγητές, ε, καθώς ε, και τα μέλη της Επιτροπής. Ε, θα πρέπει να επιμείνουμε στην εφαρμογή του γράφων αυτού επίσης. Ευχαριστώ κυρία Οβίρ. Δίνω το λόγο στην κυρία Νικολάη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την εκτίμησή μου για την έκθεση αυτή και να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Η μία είναι σημαντική, η άλλη κάπως λιγότερο. Το άρθρο 11, όπου η συγγήτρια καλεί τα κράτη-μέλη να στηρίξουν ε, ε, ευέλικτα μέτρα όσον αφορά τις ε, προσλήψεις, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια παράδοση σε αυτές τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν να κάνουν με τα δύο φύλλα. Η θέση μου είναι ότι ο λόγος που βλέπουμε αύξηση στο χάσμα απολαβών ανδρών και γυναικών είναι ότι τέτοιες συστάσεις ε, έχουν οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα. Η μεγάλη πλειοψηφία των εργοδοτών προτιμούν τις ευέλικτες συμβάσεις εργασίας και με τη χρήση αυτών των ε, συμβάσεων είναι δυνατόν να διατηρήσει κανείς το χάσμα, στις, τη διαφορά στις πληρωμές ε, στους μισθούς ατρών και γυναικών. Πιστεύω λοιπόν ότι η σύμβαση ορίστου του χρόνου θα πρέπει να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση και όχι και να μην είναι αυτές οι ευέλικτες συμβάσεις, γιατί αυτές αποτελούν την αιτία για το χάσμα, για την ψαλίδα στις πληρωμές. Θα πρέπει λοιπόν να προτιμούνται οι μόνιμες συμβάσεις και θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι οι ευέλικτες συμβάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προωθηθούν και να μονιμοποιηθούν οι διαφορές στους μισθούς ανδρών και γυναικών. Δεύτερη παρατήρηση που έχει να κάνει με την ανάγκη των κρατών μελών να παρακολουθούν συνεχώς ε, τα αποτελέσματα της διάκρισης. Μιλάμε εδώ για ένα κοινωνικό φαινόμενο. Δεν μιλάμε απλά για διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα. Πρόκειται για κοινωνικό φαινόμενο με τεράστιες συνέπειες για τα επόμενα 10 ή 20 χρόνια εάν δεν καταφέρουμε να λάβουμε προληπτικά μέτρα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε σαφείς νομοθετικές λύσεις οι οποίες να ανακουφίσουν το πρόβλημα, αλλιώς η τάση αυτή θα συνεχιστεί, η αγορά εργασίας θα συνεχίσει να είναι στρεβλωμένη και μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν βράχη πρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη προσέγγιση για το θέμα αυτό, όχι όμως μακροπρόθεσμη. Αυτό δεν είναι καλό. Μήπως θα πρέπει να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να επιτρέψουν τη συγκέντρωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, διότι στις ηλικίε 50 ε, με 65 ετών, λόγω στις ε, δυνατότητες της τεχνολογίας, οι γυναίκες μπορούν να είναι ιδιαίτερα διαστήριες ε, στην αγορά εργασίας τελευταία παρατήρηση αφορά την οστεοπόρωση. Είναι μια ασθένεια ε, την οποία αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες. Αυτή μπορεί να θεωρηθεί και επαγγελματική ασθένεια, διότι μπορεί να προκληθεί από τις συνθήκες εργασίας. Λίγα έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο βαθμό που είναι δυνατόν ίσως θα έπρεπε να αναφέρουμε την ανάγκη μέτρων για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Ε, ευχαριστώ. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Σέσκοβα. Μετά θα ακούσουμε την Κομισιόν. Πρώτα η κυρία Σέσκοβα, παρακαλώ. Eh, ευχαριστώ πολύ, κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μερικά σχόλια, καταρχήν για το σημείο 12 και μετά 24. θα ήθελα κυρίως να αναφερθώ στο θέμα των αδειών που αναφέρει το σημείο 12 και μετά το θέμα των κατωτάτων μισθών στην Ευρώπη που αναφέρει το σημείο 24. Χρειάζεται εδώ να γίνει κάποια ενημέρωση, με συγχωρείτε αν έχει ήδη υποθεί αυτό γιατί δεν ήρθα από την αρχή, ήμουν σε άλλη επιτροπή. Πρέπει να δούμε ποιος θα ωφεληθεί από τις άδειες μεταποδοχών γιατί οι εργοδότες χρειάζεται να αντικαταστήσουν τους αδιούχους από άλλους. Και όταν υπάρχει οικονομική κρίση όπως η σημερινή, είναι πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο και δύσκολο είναι να ζητήσουμε από τους εργοδότες ή από το κράτος να χρηματοδοτήσουν τις άδειες που πρέπει βέβαια κανονικά να έχουν οι εργαζόμενοι για να φροντίσουν μέλη της οικογένειάς τους. Θα σας πω τι συμβαίνει στην Τσεχία. Φυσικά πληρώνονται οι γονικές άδειες, αλλά υπάρχουν και, άλλες, και άλλα επιδόματα, κοινωνικά, οικογενειακά κτλ. Και εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι επίδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης που είναι απαραίτητη και δίκαια. Δεν αφορά μόνο την περίθαλψη των παιδιών, αλλά και άλλα μέλη της οικογένειας και άλλων μελών της οικογένειας όποτε χρειάζεται να τύχουν κάποια ιδιαίτερη φροντίδας. Ελπίζω αυτό να χρησιμοποιείται, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από γυναίκες και από άντρες, αν και θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι περισσότερες είναι μάλλον οι γυναίκες που το κάνουν αυτό. Για να μην βάλουμε τις γυναίκες σε πρωτεύουσα θέση αποκλειστικά. Το άλλο θέμα τώρα για τις συνταξιοδοτήσεις. Δίκαιο είναι και αυτό, αλλά θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω ποια συνάδελφος ακριβώς το είπε, ότι η περίοδος κατά την οποία μία γυναίκα αναγκάζεται να φροντίσει τα παιδιά της επηρεάζει τελικά αρνητικά το, τη σύνταξή της. Εγώ πήρα πληροφορίες για την Τσεχία και είδα ότι η σύνταξη υπολογίζεται για ολόκληρη την ε, εργασιακή ζωή και η περίοδος κατά την οποία η γυναίκα εγκαταλείπει τη δουλειά της για να φροντίσει τα παιδιά της συμπεριλαμβάνεται, συνυπολογίζεται. Ίσως πρέπει να το ξανασκεφτούμε γιατί δεν θα ήθελα να θεωρηθεί ότι τα πράγματα λειτουργούν χειρότερα από ό,τι πράγματι είναι. Άρα θεωρήστε λοιπόν αυτά που λέω ως υποδείγματα βέλτιστης πρακτικής. Και κάτι ακόμα που δεν αφορά τα χρηματικά στο σημείο 15 ευχαριστώ την εισηγήτρια που συμπεριέλαβε μία φράση για τις υπηρεσίες ε, εξυπηρέτησης κατοίκων όσο το δυνατόν μακρύτερης. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι η γενικότερη τάση που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ την εισηγήτρια που συμπεριέλαβε αυτή τη φράση που ήταν δική μου έμπνευσης και μετά υπάρχει και το 16 για τις οικογενειακές βοηθούς ή την, οικογενειακή, την περίθαλψη κατοίκων. Στην Τσεχία πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί θεωρούνται μη επαγγελματίες. Εγώ θα προτιμούσα να τους θεωρήσουμε επαγγελματίες. Γιατί ποιος θα αποφασίσει με ποιο συμβόλαιο γίνεται αυτή η απασχόληση ή αν έχουν δίπλωμα. Και πάλι φέρνω το παράδειγμα της Τσεχίας. Υπάρχει δυνατότητα να πάρει κανείς μια επαγγελματική άδεια για οικογενειακή ή προσωπική βοήθεια. Και οι άνθρωποι αυτοί πληρώνουν και φόρους και την κοινωνική ασφάλιση. Και οι ίδιοι αποφασίζουν σε πόσους θέλουν να χορηγήσουν τις υπηρεσίες τους. Είναι επαγγελματίες. Δεν θα ήταν το σωστότερο να αφαιθούν χωρίς καμία επαγγελματική κάλυψη αυτοί οι άνθρωποι. Και ένα τελευταίο, ένα τελευταίο που αφορά το 23. Εδώ νομίζω ότι σίγουρα είναι δυνατόν οι ηλικιωμένοι να μην γνωρίζουν ακριβώς τα δικαιώματα που ισχύουν για αυτούς ως προς τη δυνατότητα να τους χορηγηθεί βοήθεια κτλ. Εδώ λέει οι κυλιωμένες γυναίκες. Δεν νομίζω όμως ότι πρόκειται μόνο για γυναίκες. Νομίζω ότι μπορεί κάλλιστα να πρόκειται και για ηλικιωμένους. Ξέρω βέβαια ότι η ρόλος της δικής μας επιτροπής είναι κυρίως να ασχολείται με τις γυναίκες, αλλά παρόλα αυτά για το θέμα που φύγουμε εδώ το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και τελείωσα. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα η Κομισιόν. Ορίστε κύριε μου. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι με το θέμα αυτό ασχολείται συνάδελφος από άλλη μονάδα. Θα ευχαριστώ το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για ε, το σχέδιο έκθεσης πρωτοβουλίας ε, που βρίσκουμε ότι ήδη είναι πολύ ανεπτυγμένο. Ε, ιδιαίτερα εκτιμούμε την διατομεακή προσέγγιση διότι είναι θέμα που αφορά την απασχόληση, την υγεία της συντάξης και άλλα θέματα τα οποία ανέφεραν ήδη οι βουλευτές. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τα σημεια 2023 2023-2024. οσον αφορά το 2024, πράγματι η Επιτροπή ήδη έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλειών στον τομέα της ηλικίωσης της γύρανσης. Ετοιμάζουμε την πρόταση για το 2012 που θα είναι το ευρωπαϊκό έτος ε, ε, δραστηριότητας ε, κατά την τρίτη ηλικία και της αλληλεγγύης ανάμεσα στις ηλικίε. Θα έχουμε έγγραφο σχετικά με τις συντάξεις, το οποίο θα αναφέρεται και στην άτυπη φροντίδα και άλλα θέματα. Ίσως στο σημείο αυτό να υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν είναι πολύ σαφές. Αναφέρεται η παραβίαση των δικαιωμάτων των ε, ανθρώπων αυτών ε, που συνδέεται με το σημείο 23 το σχέδιο δράσης που εφαρμόζει το πρόγραμμα στη Στοχόλμη ε, τονίζει ότι ο χάρτης θεμελιωτών δικαιωμάτων θα πρέπει να αποτελεί την πηξίδα για όλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις πολιτικές. Στον στο πλαίσιο αυτό η Κομισιόν θα παρουσιάσει εντό του έτου σε μια ανακοίνωση για την πολιτική θεμελιωδών δικαιωμάτων και μια στρατηγική που θα διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του χάρτη. Στο πλαίσιο αυτό η Κομισιόν θα υιοθετεί ετήσιε εκθέσει που θα παρακολουθούν τι ε, εξελίξει όσον αφορά την εφαρμογή του χάρτη. Όσον αφορά το σημείο 24, για την Κομισιόν δεν είναι σαφές όταν μιλάμε για οδηγία βασικών υπηρεσιών, ε, τι εννοούμε, εννοούμε υπηρεσίες σε γενικού ενδιαφέροντος. Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήδη ισχύουν λαμβάνουν υπόψη τις ε, ιδιαιτερότητες της τρίτης ηλικία και δεν θα ε, χρειαστεί να ε, δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή οδηγία ε, για τις βασικές υπηρεσίες. Ωστόσο μπορεί να απαιτηθεί προσαρμογή των ισχυουσών των κανόνων που ισχύουν και τέλος μια διευκρίνηση όσον αφορά το δικαίωμα σε ένα βασικό εισόδημα η Κομισιόν ε, στην ε, διαβούλευση που έγινε σε δύο στάδια που έγινε πριν την ε, ανακοίνωση για την ενεργό συμμετοχή. Τονίζει ότι η διασφάλιση βασικού εισοδήματο είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας και ότι γι' αυτό δεν ενδείκνεται παρέμβαση της Επιτροπής. Γι' αυτό η Επιτροπή δεν πρότεινε οδηγία για ε, προγράμματα βασικού εισοδήματος, ελάχιστο εισοδήματος. Και ούτε προτίθεται για τον λόγο αυτό να υποβάλει σχετική πρόταση. Αυτά ήθελα να πω και θα ήθελα να επαναλάβω τις ευχαριστίες μας για την προσέγγιση αυτή που ήδη έχει αναπτυχθεί στην έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στην κυρία Πιετικέινεν που είναι η συγγήτρια για να κλείσει τη συζήτηση. Να σας θυμίσω ότι έχουμε άλλες δύο εκθέσεις. Ε, παρακαλώ κυρία Πιετικέινεν. Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να είμαι συντομότατη. Ευχαριστώ και την Κομισιόν και τους συναδέλφους Είμαι σίγουρη ότι θα ωφεληθεί η έκθεση από όλα όσα ακούστηκαν. Ας μην επισέλθω σε λεπτομέρειες όμως. Τέσσερις ερωτήσεις μου απευθύνθηκαν. Πρώτον, για το σημείο 5 σχετικά με την οδηγία ίσης μεταχείρισης. Θα ακολουθήσω ακριβώς αυτά που λέει η οδηγία για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας κλπ. Μετά, για το βασικό εισόδημα, κατώτατο εισόδημα, γνωρίζω καλά ποια είναι η κατάσταση του προβλήματος μεταξύ Κομισιών και Συμβουλίου και ακόμη σκέφτομαι αν πρέπει να τεθεί πολιτικά το πρόβλημα ή όχι. Γιατί οποιαδήποτε διατύπωση και να χρησιμοποιήσουμε θα χρησιμοποιηθεί μετά από τα κράτη-μέλη. Μετά για τις υπηρεσίες κοινή ωφελία. Ίσως εδώ να είναι κακή διατύπωση, αλλά κατ' εμέ εδώ εννοούνται ορισμένες υπηρεσίες που είναι ουσιώδεις για πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο τις συγκοινωνίες. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια που άγιναν ως προς το 11. Και εδώ είναι πολύ κακή η διατύπωση και πρέπει να την προσέξουμε γιατί η ιδέα που ήθελα να εκφράσω δεν ήταν να εργάζονται περισσότερο οι γυναίκες που έχουν ήδη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Γιατί αν δεν έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται έστω και μερικώς, επειδή αφροντίζουν τα παιδιά τους ή οι γονείς και τα λοιπά, τότε χειροτερεύουν τα οικονομικά τους προβλήματα και το εισόδημά τους. Αυτό ήθελα απλώ να υπάρξει ένα σύστημα στήριξης, αλλά θα το ξαναδούμε μαζί. Και θα προσέξουμε ιδιαίτερα τη διατύπωση. Τώρα για την γονική άδεια με αποδοχές. Μερικοί το συνδέουν με τη σύνταξη. Δεν είναι προφανές να συμπεριλαμβάνονται οι ώρες που εργάζονται κανείς στο σπίτι στον υπολογισμό της σύνταξης. Γιατί πολλές φορές οι γυναίκες ήδη πληρώνονται λιγότερο από τους συζύγους τους. Αλλά τα συστήματα υπολογισμού όλων αυτών διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Πώς υπολογίζεται δηλαδή το έτος ή τα, οι ώρες απασχόλησης για τη συνταξιοδότηση. Αλλά επειδή δεν είμαι ειδική για το θέμα θα ρωτήσω ειδικού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής. 29 Ιουνίου η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και υπολογίζουμε στις 14 Ιουλίου να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ θερμά την εισηγήτρια και προχωράμε απευθείας στο επόμενο θέμα που είναι οι γυναίκες εργαζόμενες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Τόμσεν για να μας κάνει μια εισαγωγή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών είδαμε μία αύξηση των επίσφαλων θέσεων εργασίας και καθόλου περίεργο οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται, υπεραντιπροσωπεύονται σε αυτές τις επισφαλείς θέσεις εργασίας ε, στην αγορά εργασία. Και πολλές φορές οι γυναίκες ως οικιακή βοηθή και ως ε, ε, εργαζόμενες σε άλλες θέσεις είναι αόρατες στην αγορά εργασίας, επίσης στο κοινωνικό έργο, στις υπηρεσίες υγείας, στις υπηρεσίες εστίασης. Σε όλε αυτές τους τομείς η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι γυναίκες. Και αφού οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στις επισφαλείς θέσει εργασίας, τα ή αρνητικές επιπτώσεις ε, τις αφορούν όλος ιδιαίτερος. Οι επισφαλείς θέσεις εργασίας όχι μόνο επιτείνουν το χάσμα μεταξύ αντρών γυναικών, αλλά είναι και εμπόδιο στη σταδιοδρομία τους και στην επαγγελματική τους εξέλιξη και παράγει φτώχεια. Γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω για τα χαρακτηριστικά των επισφαλών θέσεων εργασίας στις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές των κρατών μελών, καθώς και στη νέα ατζέντα για την ισότητα. Είναι Πρέπει να καταρρύψουμε τα φράγματα και να βελτιώσουμε την εκπαίδευση από μικρή ηλικία αναπτύσσοντας ίσως τις θέσεις εργασίας που απαιτούν γυναικείες δεξιότητες. Ζητώ από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρουν νομοθετικά μέτρα για να βάλουν ένα τέλος σε αυτές τις επισφαλείς θέσεις εργασίας που καταλαμβάνουν τόσο χαρακτηριστικά οι γυναίκες. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις η έννοια της ασφάλειας είναι ζήτημα απλώς ευελιξίας, χωρίς καμία εγγύηση ε, κοινωνικής προστασίας. Γι' αυτό τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πάρουν συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα με ελάχιστα δεσμευτικά κοινωνικά πρότυπα που θα εγγυώνται ίση πρόσβαση σε όλους τους εργαζομένους στα προνοιακά επιδόματα, ε, στα δικαιώματα υγείας και συνταξιοδότησης ανεξαρτήτως των συνθήκων εργασίας τους. Μερικές από τις πιο επισφαλείς θέσεις εργασίας καταλαμβάνονται από γυναίκες από φτωχότερε χώρες που έρχονται να εργαστούν σε μια άλλη χώρα, στην Ευρώπη, σε θέσεις που δεν απαιτούν δεξιότητες, σε καταστάσεις και σε συνθήκες που πολλές φορές είναι και παράνομες. Οι γυναίκες αυτές ε, υφίστανται καταχρήσεις, βία, ε, σεξουαλική κακοποίηση ή δεν πληρώνονται καθόλου πολλές φορές για την εργασία τους. Ε, αυτές που βρίσκονται σε αδήλωτες θέσεις εργασίας συχνά δεν μπορούν να στραφούν στις αρχές για να καταγγείλουν αυτές τις συνθήκες και τις παραβιάσεις. Πρέπει λοιπόν να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία εφαρμόζοντας ε, την ομαλοποίηση της κατάστασης των γυναικών αυτών έτσι ώστε να μπορούν να καταγγείλουν αυτές τις ε, παρατυπίες και να πάρουν και μέτρα κατά των εργοδοτών. Το θέμα της επισφαλούς απασχόλησης έχει ανακύψει σε πολλά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε πολλά πλαίσια και σε πολλά συμφραζόμενα. Ωστόσο, το θέμα των γυναικών σε επισφαλείς θέσεις εργασίας δεν έχει αντιμετωπιστεί. Χρειαζόμαστε στοχευμένη έρευνα για, την, ε, για τα έμφυλα χαρακτηριστικά των επισφαλών θέσεων εργασίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Τόμσε, να δώσω το λόγο στην κυρία σαν παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και αυτή είναι μια πολύ καλή έκθεση. Είμαστε μια πάρα πολύ ωραία επιτροπή τελικά. Κάνουμε ευφυΐες έργο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική έκθεση λοιπόν που θίγει ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα. Το παράδοξο είναι ότι τα, οι άτυπες συμβάσεις εργασίας έχουν γίνει οι πιο χαρακτηριστικές. Είναι οι πιο χαρακτηριστικές συμβάσεις εργασίας πλέον στον κόσμο. γιατί πλέον η, η κλασική σύμβαση εργασίας που όλα τα ρυθμίζει μοιάζει να είναι η εξαίρεση. Η άτυπη φύση μιας σύμβασης εργασίας ε, κατά κάποιο τρόπο προσελκύει τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Εμποδίζει τα κράτη και τους εργοδότες δεν, ε, δεν, ε, δεν επιτρέπει στους εργοδότες και στα κράτη-μέλη να προσφέρουν σωστές συνθήκες εργασίας. Νομίζω ότι οι εργοζόμενοι επιδεικνύουν πολύ μεγάλη ευελιξία στις ώρες εργασίας, στο χώρο εργασίας, δουλεύουν όσο το δυνατόν περισσότερο, προσπαθούν να συμβιβάσουν τα πράγματα με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Από την άλλη πλευρά η μερική απασχόληση είναι συχνά ευέλικτη απασχόληση και πολλές φορές οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης χρησιμοποιούνται για να καταστρατηγήσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και ιδίως των ε, γυναικών. Από αναφορές που έχουμε από τα κράτη-μέλη το υποδεικνύουν αυτό. Η άτυπη λοιπόν εργασία μπορεί να είναι κάτι καλό, αλλά μόνο μέσα στις σωστές συνθήκες. Και πολλές από τις προτάσεις της έκθεσης είναι σωστές. Μου αρέσει πολύ το σημείο 4. Το σημείο 4 πιστεύω ότι είναι ο πυρήνας της ε, έκθεσης. Η Ευρωπαϊκή Ενωσιακή Εργασιακή Νομοθεσία πρέπει να προσαρμοστεί νομίζω για να προστατεύσει τις γυναίκες. Πρέπει επίσης να το συμπεριλάβουμε αυτό στις κατευθυντήριες ε, γραμμές ε, για την απασχόληση που θα τις ψηφίσουμε αύριο. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε πολύ έντονα τη διάσταση του φίλου στις κατευθυντήριες οδηγίες για την εργασία. Και για να κλείσω, νομίζω ότι πρέπει να ε, ε, κοιτάξουμε και τους μηχανισμούς που καθιστούν δημοφιλείς τις επισφαλίστες θέσεις εργασίας, όπως ε, η υψηλή φορολόγηση των θέσεων εργασίας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, που τις κατιστά μη για, σε εκείνους, ε, μεταξύ εκείνων που προσλαμβάνουν ε, οικιακές βοηθούς, για παράδειγμα. Και έτσι πολύ συχνά οι οικιακοί εργαζόμενοι είναι παράνομα εργαζόμενοι. Δεν δηλώνονται. Νομίζω ότι και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και δεν νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε τη λύση μόνο μέσα από το συμβατικό δίκαιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κορνέλησεν. Δίνω το λόγο στην κυρία Μάισνερ και έχουμε άλλες τρεις ομιλήτριες για το θέμα αυτό, τέσσερις. Και έχουμε άλλη μία έκθεση να συζητήσουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν να είσαστε όσο γίνεται πιο σύντομες. Κυρία Μάισνερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σβένσον. Θα ήθελα καταρχήν ε, στο όνομα της ε, πολιτική ομάδα ομάδας της ΑΛΤΕ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει. Βρίσκω ότι είναι καλή η έκθεση αυτή και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα των γυναικών σε θέσει απασχόληση, διότι είναι σοβαρό πρόβλημα, είναι και πρόβλημα στα κράτη-μέλη που έχουν ευημερία. Στη Γερμανία λέμε ότι η φτώχεια είναι ε, ε, ε, γένους θηλυκού. Περισσότερες γυναίκες βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική θέση από ότι άντρες και κυρίως σε εποχές κρίσης. Το βλέπουμε αυτό. Οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από ότι άντρες. Αυτό δεν θα πρέπει να συμβαίνει οι επισφαλείς θέσεις απασχόλησης είναι αόρατες, γι' αυτό είναι σημαντικό να συζητήσουμε το θέμα. Αυτά για αρχή. Ε, ε, ε, στην έκθεση φαίνεται και πώς επηρεάζονται οι γυναίκες ανάλογα με την ηλικία τους. Αυτό το θέμα ταιριάζει πολύ καλά με την προηγούμενη έκθεση που είχαμε το ρόλο των γυναικών σε μια γυράσκουσα κοινωνία βλέπουμε ότι οι γυναίκες ε, ε, επηρεάζονται περισσότερο από την φτώχεια και ειδικά αν συνδυάσουμε τις δύο εκθέσεις. Ε, μιλήσαμε και για την έκθεση για την ψαλίδα των αμοιβών ανδρών και γυναικών. Ειδικά σε εποχές οικονομικής κρίσης ή δύσκολων συνθήκων όλα αυτά ενισχύονται. Οι διαφορές στην αμοιβή ανδρών και γυναικών οφείλεται για παράδειγμα σε διακοπή της ε, απασχόλησης, σε κάτι που οδηγεί σε ε, λιγότερη σύνταξη. Ε, σχετίζεται με το θέμα της περιορισμένης πρόσβασης σε, στην εκπαίδευση. Ένα φαινόμενο παρουσιάζεται πολύ καθαρά ότι μπορεί να είναι δύσκολο για μια γυναίκα να διατηρήσει την απασχόλησή της και την ανεξαρτησία της ε, όταν ε, έχει οικογένεια, κάτι που μπορεί να την οδηγήσει να ε, πάρει μια μισθωτή θέση εργασίας και να χάσει και εισόδημα και δυνατότητες. Ε, βλέπουμε παντού ότι χρειαζόμαστε γυναίκες ε, με ε, καλά επαγγελματικά προσόντα. Στο άρθρο 4 θα ήθελα να προσθεθεί κάτι, θα υποβάλω σχετική τροπολογία. Θα ήθελα να συμπεριληφθεί εδώ πέρα και η πρόσβαση στην εκπαίδευση. Αναφέρεται στο άρθρο 4 ότι οι γυναίκες σε επισφαλείς θέση εργασία χρειάζονται πρόσβαση στην ε, κοινωνική ασφάλιση και άλλα. Αυτό είναι σωστό. Θα πρέπει όμως να έχουν και πρόσβαση στην εκπαίδευση ώστε να μην χάσουν τις δεξιότητέ τους, αλλά να τις διατηρήσουν ώστε αργότερα να μπορέσουν να ε, ξαναβρούν ε, μια καλή θέση απασχόλησης. Ε, και επίσης αναφερόμαστε στην προσέγγιση flexicurity, την ευέλικτη ασφάλεια που θεσπίζεται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό είναι, αυτό είναι σωστό, διότι όχι μόνο για γυναίκες αλλά και για τους άντρες χρειαζόμαστε περισσότερη ε, έχουμε περισσότερη ευελιξία στις θέσεις εργασίας, αυτό δεν είναι μόνο μειονέκτημα, είναι, μπορεί να είναι και πλεονέκτημα, μπορεί για παράδειγμα να συνδυαστεί καλύτερα με την ε, οικογενειακή ζωή, αλλά η, ε, ε το flexicurity ε, περιλαμβάνει όχι μόνο ευελιξία, αλλά και ασφάλεια. Οι γυναίκες ε, συχνά ε, αναζητούν περισσότερο ασφαλείς θέσεις εργασίας λόγω της οικογένειας. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τις γυναίκες από τις επισφαλείς θέσεις Και επίσης, για παράδειγμα, όσον αφορά τις θέσεις ΟΠΕΡ, αυτό αρχικά είχε σκοπό την πολιτιστική ανταλλαγή και όχι την εκμετάλλευση. Στην πράξη όμως ε, δυστυχώς ε, καταλήγουμε σε τέτοια φαινόμενα και μετανάστριες ε, αποτελούν θύματα διπλής διάκρισης αφενός επειδή είναι γυναίκες και απετέρου επειδή είναι μετανάστες μπορεί να μην γνωρίζουν τη γλώσσα ή να μην είναι να μην έχουν καλά επαγγελματικά προσόντα. Είναι λοιπόν σημαντικό να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να επιφέρουμε αλλαγές. Αυτά. Ευχαριστώ, κυρία Σαμπό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την κυρία Τόμσον εξ ονόματος του ΕΛΚ. διότι κάλυψε το πρόβλημα πολύ, με πολύ πλήρη τρόπο. Η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας υποβάλλεται στην Επιτροπή μας τη στιγμή που η Ένωση προετοιμάζει το μέλλον της για το 2020 που το λέμε 2020. Από φέτος λοιπόν αναμένεται ήδη μία πρώτη αποτίμηση της συνθήκης της Λισαβόνας η οποία μου φαίνεται ότι δεν θα είναι πολύ θετική και θα έπρεπε να πάρουμε μαθήματα από τα λάθη μας ε, ιδιαίτερα στους τομείς όπου έχει πραγματικά αποτύχει η συνθήκη της Λισαβόνας. Μιλάμε για απασχόληση των γυναικών που δεν είναι σταθερή, αλλά το ίδιο ισχύει όλο και περισσότερο και για τους άντρες ιδίως τους πιο ευάλωτους, δηλαδή τους πτωχοτέρους. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για βράχη πρόθεσμα συμβόλαια, τότε πρέπει να διαχωρίσουμε μεταξύ των εθελοντικών τιούτων και των επιβαλωμένων που μπορεί να οφείλονται στη δύσκολη οικονομική κατάσταση ορισμένων εταιριών. Αυτά τα βραχυπρόθεσμα λοιπόν συμβόλαια μπορεί να μην είναι μια αρνητική μορφή απασχόλησης. Να μην είναι. Όταν μιλάμε λοιπόν για αυτή την μερική απασχόληση ή την προσωρινή απασχόληση, πρέπει να τη θεωρούμε σαν ευκαιρία που δίνεται στις γυναίκες, γιατί έτσι είναι πιο διαθέσιμες για άλλα πράγματα εκτός από την εργασία, όπως την απασχόληση με τα παιδιά τους. Τη μερική απασχόληση λοιπόν θα έπρεπε να εξεταστεί ως εξή Τι είναι διατεθειμένη να δώσει στις γυναίκες η κοινωνία, ιδίως στις μερικώς εργαζόμενες. Διότι πρόσφατα είδαμε ότι οι μερικώς απασχολούμενες τείνουν να είναι και από τις πτωχότερες. Άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι η κινητικότητα. Πριν από περίπου 10 χρόνια η μετακίνηση για την εργασία περιοριζόταν σε ανωτέρους υπαλλήλους που κέρδιζαν και περισσότερο. Ενώ σήμερα όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούν μετακίνηση, άρα και εδώ χρειάζεται εναρμόνιση μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματική ζωής. Επιτρέψτε μου να θέσω το εξής ερώτημα. Θέλουμε οι άντρες και οι γυναίκες να συνηθίσουν όλο και περισσότερο στις απαιτήσει της αγοράς ή θέλουμε μάλλον την αγορά να προσαρμοστεί στους ανθρώπους. Δηλαδή οι οικονομικές δραστηριότητες να τονίζουν περισσότερο, να φασίζονται περισσότερο στις ανάγκες μεταξύ άλλων των γυναικών. Μια γυναίκα θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι πιο ευάλωτη από έναν άντρα και άρα αναγκάζεται να υποστεί μια συνθήκες εργασίας που τις επιβάλλει η αγορά. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκομαι εδώ και 7 χρόνια ολόκληρα και ξέρω ότι το προσωπικό όλο και περισσότερο αρενοκρατείται Συνήθως μετανάστες είναι αυτοί που κάνουν τις βοηθητικές δουλειές στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της χειροτέρευσης της κατάστασης των γυναικών καθώς και των οικογενειών που εξαρτώνται από τέτοιου είδους κακοπληρωμένες εργασίες. Αφού πολλές φορές μιλάμε για παράνομη εργασία, μη δεδηλωμένη, και σαν γυναίκες που ασχολούνται ανεπίσημα ως οικιακές βοηθοί. Θα ήθελα να τονίσω ότι, ότι λέγω είναι γεγονός ότι αυτές οι γυναίκες που εργάζονται ως οικιακές βοηθοί δεν είναι δηλωμένες και άρα δεν θεωρούνται άνεργες ούτε και ενεργές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Θα καταθέσω μερικές δευτερεύουσες τροπολογίες, αλλά γενικά νομίζω ότι θα είμαι θετική. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, δεδομένου του πλαισίου της συζήτησης εδώ και της σχέσης του με την προηγούμενη έκθεση, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε ένα ευρύτερο κείμενο, ένα πιο γενικό λόγο, ένα γενικότερο κείμενο. Αλλά επιτρέψτε μου μερικά σχόλια πάνω σε αυτή την έκθεση, την οποία ε, να πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι το σχέδιο έκθεσης θα έπρεπε να έχει επιμείνει παραπάνω στην ανάγκη ποινικοποίηση ορισμένων ε, δραστηριοτήτων, οι οποίες γίνονται ανεκτές αυτή τη στιγμή από την κοινωνία. Μιλώ για την καταναγκαστική εργασία. Είναι ένα είδος σύγχρονου δουλείας που δυστυχώς το δεχόμαστε ή το, το ανεχόμαστε και το δεχόμαστε σε μερικές περιπτώσεις. Η καταναγκαστική εργασία δημιουργεί δια, διακρίσεις με βάση το φύλλο, οι οποίες απλώς διαιωνίζονται αν πολιτισμικά θεωρείται κάτι που μπορεί να γίνει ανεκτό. Και αυτό είναι κάτι που επιδεινώνει τη θέση των γυναικών. Δεύτερον, πιστεύω ότι η οικιακή βοηθή θα έπρεπε να έχουν ε, μεγαλύτερη θέση σε αυτή την έκθεση. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ε, οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν δύσκολες ταπεινωτικές, εξευτελιστικές ε, συνθήκες εργασίας. Τις περισσότερες φορές δεν έχουν σύμβαση εργασίας. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να παροτρινθούν, να μην ανέχονται αυτού του είδους τη δραστηριότητα, η οποία οριακά θα μπορούσε να θεωρηθεί μια μορφή καταναγκαστικής εργασίας Τρίτον, θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, μετανάστριες. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ε, μεταναστεύουν από απελπισία για να προσπαθήσουν να βρουν δουλειά σε άλλους χώρες. Η οικονομική κρίση δεν τους έχει διευκολύνει και υπάρχουν και καταστάσεις ε, στις οποίες διπλασιάζεται μάλλον ενισχύεται αυτό με εγκληματικές δραστηριότητες, με τη διακίνηση των ανθρώπινων όντων, με την μαύρη αγορά και τις δουλειές της μαύρης αγοράς. Αυξάνονται συνεχώς οι θέσεις, ε, ε, οι θέσεις εργασίας στη μαύρη αγορά και όλο και, περισσότερο, όλο και περισσότερες γυναίκες διακινούνται μεταξύ των κρατών μελών και υποχρεώνονται στο να αναλάβουν ε, κάποιες πολύ χαμηλές και χαμηλ... κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας ε, στη μαύρη αγορά εργασίας. Τα κράτη-μέλη πρέπει να κληθούν να χαράξουν πολιτικές για την αποθάρρυνση αυτών των φαινομένων, γιατί οι παράπλευρες συνέπειες αυτών των ε, φαινομένων, αυτού του φαινομένου, είναι θα είναι, θα επιφέρουν μεταξύ άλλων την αλωτρίωση της νέας γενιάς, θα οδηγήσουν σε καταστροφή της οικογένειας βασικά. Το έχουμε δει αυτό. Έχουμε δει ότι τελευταίως ε, συναντάται και το φαινόμενο αυτοκτονίας, αυξημένης αυτοκτονίας μεταξύ των παιδιών σε περιπτώσεις που οι μητέρες τους τα άφησαν ακριβώς για να δουλέψουν σε τέτοιες θέσεις εργασίας σε άλλες χώρες. Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη. Ε, Έχουν υποθεί πολλά και θα ήθελα να ρωτήσω την εισηγήτρια κάτι. Να μας εξηγήσει κάτι στο σημείο 5. Στη γαλλική μετάφραση γίνεται λόγος για ανάγκη συνδικαλισμού των γυναικών. Μα ο συνδικαλισμός είναι δικαίωμα. Δεν είναι υποχρέωση. Δεν είναι. Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι σωστή η μετάφραση ή αν εννοεί απλώς περισσότερο κοινωνικό διάλογο με γυναίκες πράγμα το οποίο θα ήταν όντως κάτι καλό. Αλλά η διατύπωση ως έχει υπονοεί ότι θα ήταν υποχρεωτικός ο συνδικαλισμός. Πράγμα που δεν μπορεί να ισχύει. Δεν ισχύουν τέτοια πράγματα στις χώρες μέλη. Πρέπει να το αναθεωρήσουμε αυτό το τελευταίο κομμάτι του πένδε. Ευχαριστώ κυρία Μωρίνη, κυρία Φιγκερέιδο. Ε, τελευταία ομιλήτρια πριν να ακούσουμε τις ε, παρατηρήσεις της Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, σίγουρα. Να σας θυμίσω ότι πέρυσι ήμουνα μεταξύ εκείνων που υπέγραψαν για ένα πιλωτικό πρόγραμμα που θα παρήχε κίνητρα για την ε, αλλαγή από επισφαλής θέσεις εργασίας σε θέσεις εργασίας με δικαιώματα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας αναφέρει να μας ενημερώσει για το τι έχει γίνει. Θα έπρεπε ήδη να μας είχε ενημερώσει. Ε, ε, σε αυτή την εποχή που οι επισφαλείς στη θέση εργασίας πολλαπλασιάζονται όλο και περισσότερο. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το 75% των νέων θέσεων εργασίας είναι επισφαλείς θέσεις εργασίας. Και σε μερικές χώρες οι γυναίκες απαρτίζουν το 90% των εργαζομένων σε αυτές τις θέσεις εργασίας. Ελάχιστες ε, θέσεις εργασίας δημιουργούνται και προκύπτουν για τις γυναίκες και οι περισσότερες από αυτές, η συντριπτική πλειοψηφία τους, είναι ανασφαλείς θέσεις εργασίας, σαν τα μανιτάρια πολλαπλασιάζονται. Η νομοθεσία στον τομέα αυτό έχει χειροτερεύσει τα πράγματα. Έχει χειροτερεύσει την κατάσταση. Τουλάχιστον στη δική μου χώρα ισχύει αυτό. Στο σημείο 4 η συνάδελφος ε, φέσει την προσοχή στις ε, διάφορες οδηγίες οι οποίες πιστεύω ότι δεν ε, λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε, να εξετάσουμε πιο προσεκτικά τα πρακτορία έβρεσης ε, θέσεων μερικής απασχόλησης. Και κάτι άλλο που ανέφερα στο παρελθόν και θα το αναφέρω και πάλι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα στη δική μου χώρα. Η νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και ιδίως των δικαιωμάτων των μητέρων υπονομεύονται έτσι ώστε να προάγονται οι μισθοί της πείνας. 450 ευρώ το μήνα. Είναι ένας κατώτατος μισθός. Αυτός είναι μισθός φτώχειας, ο οποίος μάλιστα υποβάλλεται και σε φορολογία. Για πώς θα ζήσει κανείς με έναν τέτοιον μισθό. Ε, μένεις με 220 ευρώ, πώς θα ζήσεις και θα διατηρήσεις και θα ζήσεις και την οικογένειά σου. Τα δικαιώματα των γυναικών παρά την νομοθεσία υπονομεύονται, υποσκάπτονται. Και για να και για να τις διατηρήσουν, για να τις κρατήσουν στην ε, απασχόληση, τους δίνουν ελάχιστα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία βοήθεια όσο αφορά τα ιατρικά τους ραντεβού ή τις ιατρικές τους εξετάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε θέση. Ε, μπορούμε να είμαστε υπέροχοι στα λόγια και στα χαρτιά, αλλά σας έδωσα αυτό το παράδειγμα από την Πορτογαλία. Καθόλου δεν βοηθούμε τα δικαιώματα των γυναικών με τέτοιες θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τη θέση της Κομισιόν. Τώρα δώσω το λόγο στον κύριο Παπόλα από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Για την ε, σημαντική αυτή έκθεση και το σημαντικό και το ενδιαφέρον αυτό ζήτημα. Η κρίση αυτή ήταν πολύ πιο ισχυρή από προηγούμενες οικονομικές κρίσεις και βλέπουμε να υπάρχει αυξημένη επιρροή στην ε, απασχόληση των γυναικών. Περισσότερο από ό,τι σε παλαιότερες υφέσεις στοιχεία της Κομισιόν δείχνουν ότι οι επιπτώσεις στην ανεργία ανδρών και γυναικών είναι ε, όμοιες. Οι γυναίκες ε, όμως είναι πιο πιθανό να εργάζονται σε πιο επισφαλείς ε, θέσεις εργασίας με χαμηλότερους, με χαμηλότερη αμοιβή. Αυτό λοιπόν ε, είναι ένα θέμα που επηρεάζει την ε, ισότητα των δύο φύλων. Η Κομισιόν γνωρίζει τα γεγονότα αυτά και το τονίζει αυτό στην τελευταία τη ετήσια έκθεση για την ισότητα των φύλων. Στην έκθεση αυτή η Κομισιόν τονίζει ότι η ισότητα των φύλων είναι ζωτική σημασία για να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση του στόχου οικονομική και κοινωνική συνοχή και ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία δεν συμβάλλει απλά στην οικονομική ανεξαρτησία του, αλλά είναι και το καλύτερο χέγγιο κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η Κομισιόν ε, στις 5 ε, Μαρτίου υιοθέτησε τον χάρτη των γυναικών που αποτελεί πολιτική δέσμευση της Κομισιόν το να ε, προωθήσει την ισότητα των δύο φύλων. Θα μεταφραστεί αυτό σε μια νέα στρατηγική για την ισότητα ανδρών και γυναικών που θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της επόμενης πενταετίας. Από τι πέντε προτεραιότητε του χάρτη είναι η οικονομική ανεξαρτησία. Δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα ε, αντρών και γυναικών αν δεν υπάρχει ε, η οικονομική ισότητα και ανεξαρτησία. Γι' αυτό πρέπει να προωθήσουμε τι γυναίκε στην αγορά εργασία. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ε, στις ε, γυναίκες ε, που αποτελούν θύματα και άλλων ειδών διάκρισης όπως είναι οι μετανάστριες. Επίσης θα πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα των θέσεων απασχόλησης των γυναικών διότι υπεραντιπροσπεύονται στις επισφαλείς θέσεις και στις ε, θέσει μερικής απασχόλησης. Άλλο σημαντικό θέμα το οποίο αναφέρεται στην έκθεση είναι η ανάγκη ε, ίσης αμοιβή ε, για εργασία ίσης αξια Αυτό αποτελεί προτεραιότητα του χάρτη. Μάλιστα, οι γυναίκε αντιμετωπίζουν πολλέ ανισότητες στην αγορά εργασίας και οι συνέπειε αυτών είναι η ψαλίδα στι αμοιβέ που σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat ανέρχεται σε 17,8%. Η Κομισιόν θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα, νομοθετικά και μη, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό και μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους θα εξετάσει τις δυνατότητες για να βελτιώσει το νομικό ε, ε, δίκτυο για την ε, ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Άλλο μέσο είναι η πληροφοριακή εκστρατεία που ξεκίνησε το 2009 και που θα συνεχιστεί και φέτος. Είναι σημαντικό αυτό, διότι βασικό στόχος της εξαρτίας αυτής είναι να προκαλέσει ευαισθητοποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών ε, που εργάζονται. Η Κομισιόν επίσης θα εξετάσει τη δυνατότητα βελτίωσης της Κομισιόν σε, ε, όσον αφορά άλλους ε, τύπους άδειας που σχετίζονται με την οικογένεια, όπως είναι η γονική άδεια και η άδεια κοίησης. Επίσης, για να απαντήσω σε ένα από τα τελευταία σημεία του σχεδίου έκθεσης, ε, το δίκτυο της Κομισιόν Επιρογνωμόνων ε, θα παρουσιάσει στο τέλος της ε, χρονιάς. Ε, ανακοίνωση για τις επισφαλείς θέσεις εργασίας με, με ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα των δύο φύλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τόμψεν. Θέλετε να κλείσετε τη συζήτηση σύντομα, διότι έχουμε άλλη μια έκθεση. Παρακαλώ κύριε Τόμψεν Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη να ευχαριστήσω. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για όσα είπαν και τη συμβολή τους και θα απαντήσω τώρα σε μερικές από τις ερωτήσεις που έθεσαν. Κάτι που για μένα είναι σημαντικό, καταρχήν είπε η κυρία Ζαμπόρσκα, τι έχει να προσφέρει η κοινωνία στις μερικώς απασχολούμενες όταν κανείς εθελοντικά απασχολείται μερικώς δεν έχει επαρκές εισόδημα. Και αυτό σημαίνει γίνεται επειδή είστε παντρεμένοι και εξυπηρετείτε τον σύζυγο που κερδίζει τον κυρίως μισθό. Βλέπουμε όμως σήμερα πολύ μεγάλο αριθμό διαζυγίων στην Ευρώπη. Μερικοί αναλαμβάνουν τον κίνδυνο και λένε εντάξει θα εργάζομαι μερικός, θα καθαρίζω το σπίτι και ο άντρας θα φέρνει τα λεφτά. Ο άντρα όμω φεύγει, πάει στη δουλειά και πολλές φορές δουλεύει περισσότερο γιατί η γυναίκα είναι στο σπίτι και στη δουλειά έχει μια συνάδελφο που δουλεύει και αυτή και πληρώνει φόρους σαν τον άντρα και όταν πάει στο σπίτι κάνει και αυτή όλη τη δουλειά. Οι, δικοί της φόροι λοιπόν θα έπρεπε να μεταφερθούν στην ε, μερικώς απασχολούμενη και έτσι θα είναι πιο ίση στην αγορά εργασίας γιατί αυτός δεν θα χρειάζεται να κάνει τα ίδια στο σπίτι όσο εκείνη, όπως εκείνη. Εγώ δεν είμαι υπέρ της υποστήριξης των εθελοντικός μερικώς αποσχολουμένων. Βέβαια όταν δεν μπορούν να έχουν μία πλήρη θέση οι γυναίκες αναγκάζονται να πάρουν γυναίκες. Φυσικά δεν εννοούμε υποχρεωτικό συνδικαλισμό. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου παραδοσιακά υπάρχει κοινωνικός διάλογος με τα συνδικάτα, αλλά όχι υποχρεωτικά. Τώρα για την υποχρεωτική εργασία δεν είναι αυτό το θέμα της έκθεσης. Είναι κάτι που θα έπρεπε να το βάλουμε στην έκθεση για το δουλεμπόριο, αλλά όχι εδώ. Βλέπω βέβαια ότι στα γαλλικά ειδικά και σε άλλες αγορές εργασίας υπάρχει πολύ χαμηλός βαθμός συνδικαλισμού. Αλλά υπάρχουν μέσα για κοινωνικό διάλογο στις σκανδιναβικές χώρες ο διάλογος γίνεται μόνο μέσω των συνδικάτων. Εντάξει θα το διορθώσω αυτό για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Δεν θα σας απασχολήσω άλλο. Ευχαριστώ κυρία Τόμσεν. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 29 Ιουνίου. Ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή μας 28-29 Σεπτεμβρίου. Και λίγο χρόνο έχουμε για την τελευταία έκθεση στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Πρόκειται για γνωμοδότηση για την ε, Επιτροπή Απασχόλησης ε, που έχει να κάνει με τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Να δώσω το λόγο στην κυρία Μπάουερ που είναι η συγγήτριά μας. Παρακαλώ πολύ. Νομίζω ότι μπορώ να είμαι πάρα πολύ σύντομη γιατί ήδη συζητήσαμε σήμερα το απόγευμα καλύψαμε τα βασικά ζητήματα στην έκθεση της κυρίας ε, Πέτι Κέινεν. Ε, παρόμοια είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν. Ε, εδώ πρόκειται για μία γνωμοδότηση, η οποία προετοιμάστηκε μαζί με την έκθεση Thomas Manns και η Επιτροπή Απασχόλησης ασχολείται με αυτό. Η βασική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι οι εντάσεις που ανακύπτουν μεταξύ των γενεών. Οι εντάσεις αυτές κορυφώνονται πολλές φορές και εδώ πρέπει να εξετάσουμε τους διαθέσιμους πόρους μας, οι οποίοι θα μειωθούν στο μέλλον κατά πάσα πιθανότητα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι κάτι που θα χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο, γιατί οι γενναίες χρειάζονται η μία την άλλη. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Είναι προφανές ότι είναι διαφορετικά τα προβλήματα ανάλογα με το σε ποια γενιά ανήκει κανείς. Αλλά όσο οι νεότεροι αλλά και οι γυρεότεροι ε, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αυξήσει τα όρια της απασχόλησης τα επόμενα χρόνια. Χωρίς ε, μεγάλες προσπάθειες ε, δεν είναι δυνατόν να εναρμονιστεί ο εργοσιακός με τον οικογενειακό βίο και χωρίς μια τέτοια αρμονία δεν θα είναι δυνατό να μειωθούν οι εντάσεις. Είναι αδύνατο να μειωθούν οι εντάσεις σε μια τέτοια κατάσταση. Πολλά διακυβεύονται. Μιλούμε για διακρίσεις κατά των γυναικών και όλοι έχουμε βιώσει αυτές τις διακρίσεις, αλλά αυτό το καλύψαμε σήμερα το απόγευμα. Εδώ θα ήθελα να τονίσω όλος ιδιαίτερος κάτι που ανέφερα σε σχέση και με την Επιτροπή της κυρίας Πετικάινεν και συγκεκριμένα το γεγονός ότι υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό. Τεράστιο δυναμικό το οποίο αφήνεται ανεκμετάλλευτο. Ξέρουμε ότι η διαβίου μάθηση είναι κάτι που δεν πρέπει να τελειώνει στην ηλικία των 40. Πρόσβαση σε αυτό πρέπει να έχουν και οι άνθρωποι άνω των 40. Δεν θα έπρεπε οι παλαιότερες γενναίες να μην έχουν πρόσβαση στην διαβίου μάθηση. Ευχαριστώ κυρία Πάουερ, Η κυρία Κορνέλη, ε, παρακαλώ σύντομα για να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Συμφωνώ απόλυτα ότι μιλήσαμε για, ήδη για τις γυναίκες ε, σε μια γυράσκουσα κοινωνία με την έκθεση ποιατικά. Είναι, υπάρχει σημαντική επικάλυψη ανάμεσα στις δύο αυτές προτάσεις. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε τις προτάσεις αυτές και στην έκθεση του Τόμας Μάν της Επιτροπής Απασχόλησης. Είμαι επίσης και όδηση συγγήτρια στην Επιτροπή Απασχόλησης για την έκθεση αυτή και ε, μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνεται πολύ το θέμα των ε, φύλων. Θα πρέπει να καταβάλουμε σημαντική προσπάθεια ώστε να συμπεριληφθεί η διάσταση της ισότητας των φύλων, ώστε η Επιτροπή Απασχόλησης να μπορέσει να λάβει υπόψη της ε, τη διάσταση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κώστα, μια σύντομη παρατήρηση παρακαλώ. Συμφωνώ με τις ανησυχίες της συναδέλφου Μπάουερ. Πραγματικά έλειπε λίγο αυτό στην ε, έκθεση Τόμας Μαν και θεωρώ δίκαιο να τονίσω αυτό το ζήτημα σε σχέση με τις γυράσκουσες γυναίκες, αλλά και το σημείο για τη διαβίου μάθηση πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Θα έπρεπε να εντάξουμε εδώ επίσης τη διπλή ευθύνη που έχουν οι γυναίκες και οι μητέρες στο πλαίσιο της οικογένειας, έτσι ώστε η οικογένεια να μπορεί να απορροφά τους, τους κραδασμούς σε ό,τι άλλο δεν λειτουργεί στην κοινωνία. Έτσι νομίζω προάγεται η συμφιλίωση και η στήριξη των μελών των οικογενειών. Πρέπει επίσης να κάνουμε ουσιαστική αναφορά στις πολιτικές, σε διάφορες πολιτικές, τη φορολογική πολιτική, ε, την πολιτική στέγασης, να αναφέρουμε όλες εκείνες τις πολιτικές οι οποίες συμβάλλουν σε μια εξισορρόπηση του προνοιακού συστήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ το λόγο, κυρία Μωρίν, παρακαλώ. Euh, Κάτι πολύ σύντομο. Η εργασία της κυρίας Μπάουρ είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά υπάρχει ένα σημείο το οποίο δεν αναφέρεται καθόλου. Δηλαδή, σήμερα οι γενιές των γιαγιάδων και παππούδων παίζουν ένα νέο ρόλο ως προς τα παιδιά και την οικογένεια και στη σχέση μεταξύ των γενεών δεν πρέπει να βλέπουμε απλώς την αλληλεγγύη τους ή των νεωτέρων προς τους ε, γυρεότερους, αλλά επίσης και την αλληλεγγύη των γυρεότερων προς τα παιδιά. Όλες οι μελέτες σήμερα δείχνουν ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ εγγονιών και παππούδων ή γιαγιάδων και η αλληλεγγύη, η ουσιώδης αλληλεγγύη, σε αυτό το επίπεδο τίθεται. Θα ήθελα λοιπόν αν συμφωνεί και η κυρία Μπάουερ να το συμπεριλάβουμε και αυτό γιατί είναι μια μεγάλη αλλαγή στην κοινωνία. Ε, ε, Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Επιτροπή, ο κύριος Ισκόφσκι. Um, thank you very much. Um, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα αναφέρω με ένα πάρα πολύ σύντομο σχόλιο. Ποια είναι τα σχέδιά μας ε, για την ε, γύρενση του πληθυσμού, για την προαγωγή της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία μας. υποστηρίχθηκε από όλο το σώμα της Επιτροπής, θα διέλθει από το στάδιο της διαβούλευσης δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα ονομαστεί, ποιον τίτλο ακριβώς θα έχει ε, η πρωτοβουλία αυτή, αλλά θα συμπεριλαμβάνει τους όρους γύρενση του πληθυσμού και αλληλεγγύη μεταξύ των γενναιών. Κάποια σχόλια. Ε, καταρχήν το άρθρο 25 και την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Οικογένειες. Η διατύπωση από δεδειγμένες καλές πρακτικές ίσως είναι πολύ περιοριστική. Καταρχήν υποδηλώνει ότι υπάρχει κάτι σαν μια γενική κατεύθυνση προς την οποία προσανατολίζεται η ευρωπαϊκή οικογένεια και ότι κάποιες πρακτικές μπορούν να αποδεδειγμένα να βοηθήσουν την κατάσταση ενώ άλλε όχι. Από τη συζήτηση που είχαμε σήμερα ε, κατάλαβα ότι εξαρτάται πολύ από το κάθε κράτος μέλος καθώς και με τους υπεύθυνους της οικογενειακής πολιτικής του κάθε κράτους μέλους. Τώρα για το θέμα της μερικής απασχόλησης αυτό διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Σε μερικές χώρες είναι πολύ καλό να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες να καταλάβουν κάποιες θέσεις απασχο... περιορισμένης εργασίας, απασχόλησης ε, έστω και ως οικιακές ε, βοηθή. Σε άλλες χώρες πάλι είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες αυτές να καταλαμβάνουν θέσεις ολικής απασχόλησης και σε άλλες χώρες όπως οι κάτω χώρες προάγουν ε, περισσότερες θέσεις μερικής απασχόλησης για τους άντρες και περισσότερες θέσεις ολικής απασχόλησης για τις γυναίκες και θα μένει να αποδειχθεί ποια είναι η καλύτερη πρακτική. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερο να το συζητήσουμε ε, κατά την ανταλλαγή εμπειριών που θα έχουμε. Τώρα, στο σημείο 26 θα μπορούσε να γίνει μια αναφορά και στην τηλεεργασία ως ένα άλλο μέρος στήριξης ε, της συμφιλίωσης μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Είναι όλο και πιο σημαντικό ε, να είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι πολλής χρόνος ξοδεύεται στο, στη μετακίνηση μεταξύ της θέσης εργασίας ε, και του σπιτιού. Ε, η τηλεεργασία μπορεί να είναι ένας τρόπος παραμονής στο σπίτι και επίβλεψης και των παιδιών. Τέλος, αναφέρθηκε ότι ε, το θέμα συνδέεται με πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναλυθεί στο παρελθόν. Ε, θα ήθελα να αναφέρω ορισμένες από αυτές. Μια ενδιαφέρουσα ιδέα που νομίζω θα μπορούσε να αναπτυχθεί και σε αυτή την έκθεση ε, θύχτηκε από την κυρία Παλιαδέλη. Πρόκειται για την ενδυνάμωση των πιο ηλικιωμένων ε, και τη συμμετοχή τους στην ε, διαχείριση των ε, νοσηλευτικών θεσμών. Επίσης η κυρία Νικολάη έθιξε το θέμα της ενδοκινοτικής μετανάστευσης. Σε μερικά, σε μερικά κράτη-μέλη οι γονεί τη οικογένεια εργάζονται σε άλλο κράτο μέλο. Αυτά είναι λίγα από τα, από τα σημεία που ήθελα να θίξω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπάουερ, μια πολύ πολύ σύντομη τελική παρατη... παρέμβαση. Παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι τελείωσε ο χρόνος μας, γι' αυτό θα ήθελα απλώ να σας ευχαριστήσω για όλα σας τα σχόλια. Μία μόνο σύντομη δήλωση στα σχόλια της Ελισαβέτας θυμάμαι ότι υπάρχει το παράδειγμα ενός ουγγρικού νομοσχεδίου κατά το οποίο η γονική άδεια χορηγούνταν και για τους παπούδες και τις γιαγιάδες. Αυτό ίσως ήταν μια καλή ιδέα. Καλή. Ως παράδειγμα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ. Σας ευχαριστώ.